Dear colleagues, I wonder if you could please take your seat. Συνάδελφε, καθίστε διότι αρχίζουμε, λέει ο πρόεδρος. Please uh, be seated. Thank you. Αγαπητοί, συνάδελφοι αγαπητοί βουλευτές, καλώς ορίσατε σήμερα όλοι. Ιδίω να καλοδεχτούμε του ε, συναδελφού από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επίση, καλώ ήρθαν και οι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε αυτή την ε, παράταση τη εβδομάδα, εδώ Πέμπτη και Παρασκευή. Σα ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον μα που δείξατε για αυτή τη συνδιάσκεψη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση κατόπιν του έργου που επετέλεσαν οι ευρωβουλευτές που παρίστανται τώρα εδώ, που έλαβαν μέρος στην έρευνα της τελευταίας θητείας επίσης. Είναι ένα θέμα επίκαιρο και σημαντικό. Α, και εσείς, οι βουλευτές των Εθνικών Κοινοβούλιων, έχετε ασχοληθεί το θέμα αυτό στα κράτη-μέλη αφορά αυτή η συνάντηση τη δημοκρατική εποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή μας των ε, Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων οργανώσαμε με την ε, Πάγια Επιτροπή π και ΑΕ της ε, Βελγικής Βουλής επίσης και το πάνελ της Γερμανικής Βουλής για την κοινοβουλευτική εποπτεία αλλά επίσης και την Επιτροπή Ασφάλειας του Ιταλικού Κοινοβουλίου, οπότε πασχίσαμε τα τρία αυτά κοινοβούλια να καταφέρουμε να οργανώσουμε αυτή τη συνάντηση και μεγάλη μας ε, χαρά διαπιστώνουμε ότι έχουμε 38 βουλευτές από 17 εθνικά κοινοβούλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Νορβηγία. Επίση παρίσταται ο πρόεδρο τη Βελική Βουλή, ο κύριος Σίγφριντ Μπράκε. Επίση έχουμε 14 Πρόεδρους κοινοβουλευτικών επιτροπών και 5 αντιπρόεδρου. Πολύ επομένω σημαντική κοινοβουλευτική. Επίση, με χαρά μου, έχουμε καλωσόρισαν οι εμπειρογνώμονε από τι διάφορε χώρε, όπω επίση και οι συνάδελφοι τη Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ. Είναι επομένω πολύ σημαντικό θέμα για την κοινωνία και για του συμπολίτε μα. Οι υπηρεσίε πληροφοριών προστατεύουν τι δημοκρατικέ κοινωνίε από τι απειλέ. Αλλά βέβαια σε μια δημοκρατική κοινωνία θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία σε αυτέ τι ε, υπηρεσίε ακόμα ε, και εάν θα πρέπει να εφαρμόζονται ειδικέ διαδικασίε λόγω τη ιδιομορφία αυτών των ε, υπηρεσιών. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα είναι να δώσουμε μια συνέχεια στο ψήφισμα τη 12η Τύπου του 2014 όσον αφορά το πρόγραμμα παρακολούθηση των ΗΠΑ. Του φορεί ε, παρακολούθηση σε διάφορα κράτη-μέλη και τι επιπτώσει ε, στου ε, πολίτε. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων πρότεινε την οργάνωση μιας τέτοια συνδιάσκεψη σε σχέση με τις, ε, τους, τους φορείς εποπτείας των εθνικών Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων. Με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι έχουμε τρία κοινοβούλια καθώς και τους φορείς αυτών που δέχτηκαν να συμμετάσχουν. Είπαμε μόνο ότι έχουμε την Βελγική Βουλή, τη Γερμανική Βουλή, έχουμε την αντίστοιχη υπηρεσία και επιτροπή της Ιταλικής Βουλής. Έχουν γίνει επίσης τέτοιες συναντήσεις στο παρελθόν, σε Ρώμη, Βρυξέλλες και Βερολίνο. Ελπίζω ότι και στο μέλλον θα προχωρήσει αυτή η συνεργασία. Και τώρα δώσουμε τον λόγο στην κυρία Σολβίτα Αμπολτίνα, που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής ε, Ασφαλείας της ε, ε, Λετωνίας, του Κοινοβουλίου της Λετωνίας. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να γίνει, μια που τώρα βρισκόμαστε ε, υπό λετωνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και έχετε την σκητάλη για την εισήγησή σας. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Μωράς, κύριε και κύριοι. Είναι πραγματική μου τιμή το γεγονός ότι έχω τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτή τη διάσκεψη που αφιερώνονται στα ζητήματα που σχετίζονται με την ε, εθνική ασφάλεια των κρατών μελών. Όπως γνωρίζετε, η Λετωνία βρίσκεται στην πρώτη, φάση, ε, στην πρώτη προεδρία ε, της, ε, του Συμβουλίου. Και μια από τις προτεραιότητες που έχει ορίσει πριν από την ανάλυση Προεδρίας ήταν η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της κοινή ε, πολιτικής άμυνας και της κυβερνοασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την τρομοκρατία, τονίσαμε ότι θα ασχοληθούμε με ζητήματα τρομα, τρομοκρατίας, ριζοσπαστικοποίησης και ξένων μαχητών. Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια σειρά από απειλές από διεθνείς ομοκρατικές οργανώσεις μέχρι ε, τρομοκράτες που προσπαθούν να απειλήσουν την δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλειά μας. Η φύση της ε, ασφάλειας στην Ευρώπη έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Η Ευρώπη ε, έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα οι πράξεις της ε, Ρωσίας με την ε, προσάρτηση της ε, Κρυμαίας και την απεσταθεροποίηση της Ανατολικής Ουκρανίας δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα η ανθρώπινη τραγουδία χιλιάδων προσφύγων στην Νότια Ευρώπη καταδεικνύει ότι τα προβλήματα εντείνονται στην γειτονιά μας. Η απειλή του οργανωμένου εγκλήματος οι ε, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, τα όπλα που ε, αναπτύσσονται και οι μέθοδοι χρηματοδότησης των τρομοκρατικών οργανώσεων απαιτούν ε, οι, πληροφορίες, οι υπηρεσίες πληροφοριών να διατηρούν τις ικανότητές τους ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τις απειλές προτού υλοποιηθούν σε κάτι συγκεκριμένο. Από την εμπειρία μας ε, μπορώ να σας πω ότι από τα τροκοματικά ε, χτυπήματα στο Παρίσι, μακριά από τη Λετωνία δηλαδή, ε, ακόμη και η ασφάλεια του δικού μου λαού ε, θεωρούμε ότι έχει υπονομευθεί. Και καταφέραμε και αντιμετωπίσαμε τα, τα προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια χάρη στην διεθνή συνεργασία. Αυτό αποδεικνύει ότι όλοι αντιμετωπίζουμε τις ίδιες διεθνείς ε, απειλές και μαζί θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Οι υπηρεσίες πληροφοριών θα πρέπει να έχουν και εξουσίες και να λειτουργούν με μυστικότητα. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα των πολιτών και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η εθνική ασφάλεια. Υπάρχει λοιπόν αυτό το δίλημα ε, για την προστασία της ιδιωτικότητας και της εθνικής ασφάλειας, η οποία μπορεί να, το οποίο μπορεί να επιληθεί μόνο μέσω της δημιουργίας ε, θεσμών. Αυτοί οι θεσμοί θα πρέπει να είναι δημόσιοι, αλλά δεν μπορεί πάντοτε να λειτουργούν με πλήρη διαφάνεια. Σήμερα πιστεύω ότι οι άνθρωποι ε, είναι πιο πρόθυμοι να δίνουν ε, τα προσωπικά τους δεδομένα σε ιδιωτικούς παράγοντες, για παράδειγμα για να έχουν εκδόσει σε σούπερ μάρκετ, αλλά όταν κάποια εθνική υπηρεσία ζητά δεδομένα των πολιτών, θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να εργαστούμε ώστε να γίνει κατανοητή οι... ποιοι είναι οι κανόνες και πώς θα τηρούνται. Είμαι πεπισμένη ότι η εποπτεία και η επιτήρηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην, στο έργο των ε, υπηρεσιών πληροφοριών. Γιατί αυτές είναι σημαντικές και θα πρέπει το έργο τους να προστατευτεί. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι η εθνική ασφάλεια είναι εθνική αρμοδιότητα, θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι η ανάγκη για την αντιμετώπιση των απειλών και της αντιμετώπισης της ε, ριζοσπαστικοποίησης του 21ου αιώνα θα πρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία μας με συμμάχους και εταίρους και να απαντήσουμε με θετικό τρόπο στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις όσον αφορά τις εξουσίες που έχουν οι μυστικές μας υπηρεσίες στο έργο τους για τη διατήρηση της ε, ασφάλειάς μας σε ένα ταχαίως μεταβαλλόμενο περιβάλλον τεχνολογικό. Από την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ε, ιδιωτικότητα και η δημοκρατία ήταν πολύ σημαντική και Πιστεύω ότι σήμερα αυτό δεν έχει αλλάξει. Η ειρήνη, η σταθερότητα και η ευημερία θα είναι το πλαίσιο για να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις εν ώψη των αλλαγών που αντιμετωπίζουμε σήμερα και που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ο κόσμος χρειάζεται την Ευρώπη και είναι στο δικό μας χέρι να συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να ε, θέτουμε πάντοτε στο επίκεντρο κοινό καλό. Είμαι πεπισμένη ότι σήμερα θα ακούσουμε πολλές σημαντικές και ενδιαφέρουσες ιδέες για το πώς μέσω της στενότερης συνεργασίας μας θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την διεθνή συνεργασία. Ελπίζω να έχουμε μια επικοδομητική διάσκεψη και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, Ms. Thank you. Σας ευχαριστούμε κυρία Αμπουρτίνα. Ε, δώσατε έμφαση σε πολύ ενδιαφέροντα στήματα που θα διερευνήσουμε διεξοδικότερα. Τώρα θα αρχίσουμε το πρώτο τμήμα σε σχέση με τις, ε, τον αντίκτυπο που έχει η, η επόπτευση των υπηρεσιών πληροφοριών σε ένα ε, κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία. Θα ακούσουμε τον κύριο Σίκφριτ Πράγκε που είναι ο πρόεδρος ε, ε, της αντίστοιχης επιτροπής ε, στην, ε, στο Βελγικό Κοινοβούλιο θα ήθελα προτού γίνει η παρέμβαση του κ. Μπράκη να κάνουμε μια παρουσίαση της σημερινής συζήτησης. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συμμετέχοντες να δηλώνουν επιθυμία τους να μιλήσουν στην αρχή κάθε τμήματος συζήτησης ή κάθε εργαστηρίου. Υπάρχουν ε, καρτελάκια διαφορετικού χρώματος για κάθε τμήμα της συνεδρίασης από ό,τι φαίνεται. Οπότε έχετε για την τωρινή σύνοδο ε, μία κάρτα για το ε, χρώματος ροζ, μπλε για το πρώτο εργαστήριο και το καθεξής. Για τα μέλη του, για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν χρειάζονται αυτές οι κάρτες, μπορείτε απλώς να σηκώσετε το χέρι. Οι υπόλοιποι παρακαλώ να χρησιμοποιείτε αυτά τα καρτελάκια. Ροζ χρώματος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άμα δεν θέλετε και να τα χρησιμοποιήσετε, θα δείξουμε ευελιξία. Προτού όμως ε, παρέμβετε, θα ήθελα να παρουσιάζεστε, να μας λέτε από πού είστε και το όνομά σας. Μετά από τους βασικούς ομιλητές, κάθε σύνοδου θα ακούσουμε δύο από κάθε κοινοβούλιο, από τι αρμόδιε επιτροπέ και εμβόλυμα θα ακούμε και έναν βουλευτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ο τρόπο που βρήκαμε για να έχουμε το μέγιστο αριθμό παρεμβάσεων από του αρμοδίου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ελπίζουμε να είναι ζωηρή συζήτηση και παρακαλώ δηλώστε την επιθυμία σας να μιλήσετε. Επίσης θα γίνει μια, ένα κοκτέιλ μετά την απογευματινή μας σύνοδο ακριβώς έξω από την αίθουσα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε άλλο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπράκε τώρα που θα πάρει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι ε, μας τιμά που είμαστε σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες ε, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική διάσκεψη διότι είμαι βαθύτερα πεπισμένος ότι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα και αύριο θα έχει αυξανόμενη σημασία στο άμεσο μέλλον και στο απότερο μέλλον από ό,τι φοβάμαι. Μετά την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων στο ψήφισμα της 12 Μαρτίου 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκάθαρα εξέθεσε τις ελλείψεις που υπάρχουν στη δημοκρατική ε, ποπτεία των υπηρεσιών πληροφοριών. Πρώτον, φαίνεται ότι οι εθνικοί οργανισμοί και φορείς δεν έχουν προσαρμοστεί ή όχι επαρκώς ε, στις ραγδαίες πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις τελευταία δεκαετία. Δεύτερον, η εποπτεία ασκείται ακόμη ε, σε εθνικό επίπεδο παρά την ε, αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών ε, ανάμεσα στις υπηρεσίες πληροφοριών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τρίτες χώρες και τρίτος αναφέρεται η έκθεση στο διωγούμενο χάσμα ανάμεσα στο επίπεδο της διεθνούς συνεργασίας αφενός και των περιορισμένων δυνατοτήτων υποπτίας σε εθνικό επίπεδο αφετέρου που μας οδηγεί και παραθέτω από την έκθεση σε, μια ανεπαρκή και ένα ανεπαρκή και ένα αποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή δεν είναι, είναι ζωφερή μάλλον η εικόνα ε, γενικότερα η εθνικοί φορείς ε, είναι σχολαστική και μπορώ να σας πω ως πρόεδρος της Αρμόδιας Επιτροπής ε, στο Βελγικό Κοινοβούλιο ότι η Βελγική Επιτροπή αποτίμησε και προβληματίστηκε με ιδιαίτερα ασφαλή τρόπο για τις αποκαλύψεις Snowden σε σχέση με το ρόλο δηλαδή των βελγικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ε, παρόλα αυτά, η ενισχυμένη διεθνή συνεργασία υποχρεώνει το σύστημα δημοκρατικού ελέγχου να λάβει υπόψη αυτή την εξέλιξη. Ο Χάν Μπον και ο Λόγ Σόνσον ε, πριν από λίγο καιρό, που είναι δύο εμπειρογνώμονε αναγνωρισμένοι ε, στο τομέα αυτό, αναφέρθηκαν σε πέντε χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ελέγχου. Πρώτον, πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα ένα τέτοιο φορέα από την εκτελεστική εξουσία και από τι περιουσίε πληροφοριών. Επίση, θα πρέπει να έχει την ελευθερία επιλογή των ερευνών που θέλει να διεξάγει. Τρίτον, ένα φορέα πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα διαπιστευμένα, διαβαθμισμένα συγγνώμη, έγγραφα και τι πληροφορίε και πέμπτον πρέπει να έχει επαργέ σε προσωπικό εκτεταμένο σε νομικές αρμοδιότητες και οικονομικά μέσα για να ασκήσει τα καθήκοντά του. Υποστηρίζω πλήρω αυτά τα χαρακτηριστικά, όμως είμαι πεπισμένο ότι δεδομένων των εξελίξεων, αυτές, αυτά τα πέντε χαρακτηριστικά πηχούν μόνο εν μέρει την πραγματικότητα. Και, και επίσης δεν αναφερόμαστε καθόλου στο διεθνές περιβάλλον. Στις εκτεταμένες συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο είναι ξεκάθαρο Ω προ αυτό και παραθέτω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί για αυξημένη συνεργασία ε, για την εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως για τη διασυνοριακή διάσταση και επίσης, και εξακολουθώ να παραθέτω, απευθύνει έκκληση προς τα κράτη-μέλη για να αναπτύξουν συνεργασία ανάμεσα στους εθνικούς φορείς εποπτείας. Έχουν γραφεί πολλά για αυτό το πράγμα στο παρελθόν, αλλά πρακτικές πρωτοβουλίες με την εξαίρεση κάποιων διμερών σχέσεων έχουν παραμείνει ε, στο χαρτί. Δεν έχουν εφαρμοστεί και ε, γι' αυτό και επικροτούμε την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διοργανώσει αυτή τη διάσκεψη τώρα. Θα πρέπει να πάρουν τη σκητάλη και να δεχθούν αυτή την πρωτοβουλία οι εθνικές αρχές ε, εύχομαι να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση σήμερα το πρωί. Σας ευχαριστώ. Uh, Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ήλκα Σάλμη που είναι ο Διευθυντής ε, του ε, Κέντρου Ανάλυσης Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και των Μηχανισμών Λογοδοσίας πρέπει να φύγει στις 10 που μας έχει ενημερώσει οπότε θα του δώσουμε χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχά να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ σε εσά σήμερα εδώ το πρωί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΙΝΤΣΕΝ, με συγχωρείτε, να έχει την δυνατότητα να σα παρουσιάσει το έργο μα. Γιατί πολλέ φορέ ε, υπάρχουν κάποιε παρεξηγήσει, κάποιε παρανοήσει όσον αφορά τι δραστηριότητε μα. Θα προσπαθήσω να χωρίσω την παρουσίασή μου σε τρία μέρη. Πρώτον, θα προσπαθήσω να περαγράψω τις, ε, τις ε, δραστηριότητες μας, πώς, ε, ποιο είναι το οργανόγραμμά μας και τι είδους πράγματα κάνουμε δηλαδή. Δεύτερον, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις διαφορές μεταξύ των δικών μας δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων των εθνικών μυστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασφαλείας. Και να σημειώσω ότι είμαι πρώην διευθυντή των Φιλανδικών Μυστικών Υπηρεσιών, οπότε ξέρω και ποια είναι η, η άλλη πλευρά και θεωρώ ε, δηλαδή ότι γνωρίζω ε, ποιες είναι οι σκέψεις και οι απόψεις των εθνικών υπηρεσιών. Και τρίτο θα ήθελα να πω δύο λόγια για τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την νομική βάση των δραστηριοτήτων μας. Ε, κάποια από τα πρόσφατα πορίσματα ε, στα οποία κατέληξε το Κοινοβούλιο η Κομισιόν όσον αφορά τις δραστηριότητες του ΕΣΕΝ. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να σας τα πω, γιατί ήρθα από μακριά και θα πρέπει δυστυχώς ε, στις 10.30 να έχω επιστρέψει στο γραφείο μου. Οπότε για να μπορέσετε να κάνετε και τις ερωτήσεις σας θα προσπαθήσω να μιλήσω πολύ λίγο. Λοιπόν, Είμαι Φιλανδός ε, και έχω 20 χρόνια εμπειρία στις μυστικές υπηρεσίες, οπότε νομίζω θα τα καταφέρω. Δραστηριότητες της Twinsen. Δύο βασικά πράγματα να σας πω. Πρώτα απ' όλα είμαστε τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε διεύθυνση εντός της υπηρεσίας αυτής. Έχουμε περίπου 80 υπαλλήλους από σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ακόμη κάποιες μυστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ασφαλείας που ακόμη δεν έχουν μετατάξει ε, υπάλληλό τους στην, ε, δική μας, ε, στο δικό μας κέντρο αλλά μπορώ να σας πω ότι οι περισσότερες υπηρεσίες από τα κράτη-μέλη ε, εκπροσωπούνται. και υπάρχουν άνθρωποι και από τις, από τις υπηρεσίες της Εθνικής Ασφάλειας και από τις Εθνικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Και θέλω να τονίσω από την αρχή. Εμείς δεν είμαστε οργανισμός με επιχειρησιακές δυνατότητες. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες, δεν έχουμε ε, δικαίωμα ε, να αξιοποιούμε τέτοιου είδους ε, πληροφορίες, ούτε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα. Και αυτές είναι οι βασικές μας διαφορές όταν κανείς συγκρίνει τις δικές δραστηριότητες με τις δραστηριότητες των εθνικών υπηρεσιών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και όσον αφορά το ζήτημα της εποπτείας των δικών μας δραστηριοτήτων. Όχι. 500 εκθέσεις ε, συντάξαμε πέρσι. Ε, είναι στρατηγικής φύσης, δεν έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε πληροφορίες στρατηγικού χαρακτήρα ή τακτικού χαρακτήρα. Ε, περισσότερο κοιτάμε ε, σε ποιες περιοχές ε, θα μπορούσαν ενδεχομένως να πληγούν τα συμφέροντα ή οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνο ζήτημα το οποίο εξετάζουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συνδέεται με την αντιτρομοκρατία και την κυβερνοασφάλεια και τα σχετικά ζητήματα. Η οργάνωσή μας χωριζόμαστε σε δύο τμήματα. Υπάρχει το τμήμα ανάλυσης στο οποίο εργάζονται 45 ε, υπάλληλοι των εθνικών υπηρεσιών. Υπάρχουν και κάποιοι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιοι σαν εμένα που έχουμε εμπειρία ε, από εθνικές υπηρεσίες αλλά ε, είμαι ε, υπάλληλος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προσωρινή βάση. Υπάρχει και ένα άλλο τμήμα που χωρίζονται, σε 7 υποτμήματα, 7 4 ε, περιφερειακά και 3 θεματικά. Ε, η κυρία Μογκερίνη ε, είναι αυτή στην οποία λογοδοτούμε εμείς, αλλά υποβάλλουμε τις εκθέσεις μας και σε όλους τους, ε, σε όλους τους άλλους, σε όλα τα άλλα θεσμικά όργανα, Συμβούλια, τον Πρόεδρο της Κομισιόν, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, ενημερώνουμε τις ε, ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, πάνω από 200 τέτοιες ενημερώσεις κάναμε πέρσι για διάφορα ζητήματα. Και, όπως είπα, περισσότερα, ε, συντάξαμε περισσότερες από, περισσότερα από 500 ενημερωτικά σημειώματα πέρσι. Τώρα, όσον αφορά τις πηγές, όπως είπα δεν έχουμε δικαίωμα συλλογής πληροφοριών. Οπότε στην ουσία βασιζόμαστε ε, στις πληροφορίες που λαμβάνουμε από τις ε, εθνικές υπηρεσίες. Ε, αυτό είναι το μονοπόλιο που έχουν και από αυτή την άποψη είμαστε μια, ένα κέντρο πολιτικών πληροφοριών. Λάβαμε χιλιάδες πληροφορίες πέρσι και Πρέπει να σας πω ότι τα τέσσερα χρόνια που εργόζομαι σε αυτή τη θέση ε, έχει βελτιωθεί και η ποσότητα και η ποιότητα των πληροφοριών. Υπάρχει δηλαδή μια σαφής δέσμευση των εθνικών υπηρεσιών να μας βοηθούν ε, δίνοντάς μας τις ε, πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό στοιχείο και θεωρώ, είμαι βέβαιος, ότι και η ύπατη εκπρόσωπος ε, ε συμμερίζεται την άποψη αυτή. Φυσικά βασιζόμαστε και σε δημόσια προσβάσιμες ε, πληροφορίες. Ε, το άλλο τμήμα μας ε, ε, για τις εξωτερικές σχέσεις ε, βασίζεται ακριβώς αυτό. Και όπως είπα δεν έχουμε δικαίωμα να ε, διεξάγουμε μυστικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η πρόσβασή μας αφορά μόνο πληροφορίες που είναι δημόσια προσβάσιμες. Αλλά και αυτές είναι πολύ χρήσιμες. Τρίτη πηγή για τις αξιολογήσεις μας είναι οι εκθέσεις των ε, αντιπροσωπείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν 140 τέτοιες αντιπροσωπείες και οι εκθέσεις που υποβάλλονται ε, από αυτές τις αντιπροσωπείες είναι πάρα πολύ σημαντικές για το έργο μας. Οι δικές μας εσωτερικές δυνατότητες, η δυνατότητα είναι η συνεργασία μας με το Κέντρο Διαστημικής Δράσης ε, στην Ισπανία συνεργασία που έχει αποδειχθεί ότι ήταν πολύ σημαντική και ε, το τελευταίο διάστημα με τις, με τις συγκρούσεις που υπάρχουν στα ε, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουμε συνεργασία με το EUMS που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, συνεργαζόμαστε και με, τους, ε, με, τους, ε, με τις στρατιωτικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Και αυτό είναι και επιθυμία των πελατών μας, δηλαδή να παρέχουμε και τέτοιο είδους πληροφορίες και Πιστεύω ότι μπορούμε πραγματικά να ε, συνδυάσουμε στις εκθέσεις μας αυτού του, αυτές, τις δύο κατηγορίες πληροφοριών, τις στρατιωτικές και τις πολιτικές. Λοιπόν, δεύτερο σημείο. Ποιες είναι οι διαφορές μας. Είπαμε, δεν έχουμε επιχειρησιακές δυνατότητες, δεν ε, συλλέγουμε πληροφορίες και πληροσωπικά δεδομένα. Από άποψη ιδιωτικότητας αυτό το τελευταίο σημείο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να κατανοηθεί για να καταλάβει κανείς και τον δικό μας ρόλο. Και να σας πω την αλήθεια, ακριβώς για να επιτελέσουμε εμεί το έργο μας δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδους ε, πληροφορίες, ούτε θεωρώ ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή η δική μας υπηρεσία να ε, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πολιτών. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, αυτό που κάνουμε εμείς είναι στρατηγικές έρευνες για ζητήματα που ε, ενδεχομένως να αποτελέσουν στρατηγικής ε, σημασίας θέματα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τι έχει υποθεί πρόσφατα για τις δραστηριότητε μας και υπήρξε ήδη μια αναφορά σχετικά με τις εκθέσεις για το πρόγραμμα ε, επιτήρησης του NSA όπου ο εισηγητής ήταν ο κύριος Μωράες Υπήρξε λοιπόν μια σαφής δήλωση που αφορούσε και τον ρόλο του Ίντσεν και το πώς οι δραστηριότητες του κέντρου μας θα πρέπει να παρακολουθούνται. Και να σας παραθέσω ένα σημείο από αυτή την έκθεση. Καλεί λοιπόν το HREP να ε, ε, λογοδοτεί για το ΙΝΤΣΕΝ και τις δραστηριότητες του ως τμήμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας εσωτερικής δράσης και να λογοδοτούν στα, στις αρμόδιες επιτροπές, επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διαπιστώνουν τη συμμόρφωσή τους με τις βασικές κανόνες περί ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλείται λοιπόν η Επιτροπή και οι εκπρόσωπους να υποβάλουν μια πρόταση για τη νομική βάση των δραστηριοτήτων του Ίντσον σε περίπτωση που στο μέλλον αποκτήσει ή επιχειρηθεί να αποκτήσει δικές του αρμοδιότητες συλλογής προφοριών και προσωπικών δεδομένων. Ε, είναι κάπως υποθετικό δηλαδή ότι αν οι δραστηριότητες μας αποκτήσουν ένα περισσότερο επιχειρησιακό χαρακτήρα τότε θα πρέπει να υπάρχει σαφής μηχανισμός επιτήρησης εποπτείας των δραστηριοτήτων μας. Όπως είπα, κάτι τέτοιο ε, ούτε συμβαίνει τώρα, ούτε φαίνεται να ε, συμβεί κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον. Η Κομισιόν απάντησε σε αυτή την έκθεση, επίσης, και αφορά και το ζήτημα της νομικής βάσης των δραστηριοτήτων μας. Όπως είπα, το ίντσεν είναι τμήμα της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και από αυτή την άποψη η νομική βάση των δραστηριοτήτων του ίντσεν είναι αυτή που ε, αναφέρεται στην απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής ε, Δράσης. Και ε, οι κανόνες που περιέχονται στην απόφαση αυτή αφορούν βεβαίως και το Ίντσεν, το δικό μας κέντρο. Και να αναφερθώ και σε ένα ζητήμα που πολλές φορές ανακύπτει όταν μιλώ για, τα, για τις δραστηριότητες του Ίντσεν. Έχουμε τη δυνατότητα εμείς να ελέγχουμε τις συμβολές των κρατών μελών. Πρώτον, όλες οι συμβολές έχουν εθελοντικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει δηλαδή μηχανισμός. Μπορούμε να ζητήσουμε πληροφορίες, αλλά δεν μπορούμε να αναθέσουμε να μας δοθούν κάποιες πληροφορίες. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Επίσης δεν έχουμε πρόσβαση στον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες αυτές έχουν συλλεγεί ή τι είδου συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή των πληροφοριών. Αλλά γι' αυτό είναι η αφετηρία μας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην γνώμη, στη γνώμη του το 2013 ανέφερε ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών είναι εξαίρετη σημασία στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάθε κράτος μέλος να ε, εξετάζει ή να αμφισβητεί αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς ακριβώς αυτόν τον κανόνα ακολουθούμε. Θεωρούμε δεδομένο ότι έχουν ακολουθηθεί όλοι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής και της, και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και του Διεθνούς Δικαίου. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό δηλαδή. Και μια τελευταία παρατήρηση όπως είπα, δεν έχουμε ε, μηχανισμό για την ανάθεση ζη, συλλογής πληροφοριών. Όμως μπορούμε να ζητούμε πληροφορίες. Ζητούμε εκατοντάδες, ε, εκατοντάδες τέτοια αιτήματα ετησίως και λαμβάνουμε και μεγάλο αριθμό απαντήσεων. Επίσης, πολλές φορές λαμβάνουμε πληροφορίες χωρίς να τις έχουμε ζητήσει και αυτό αποδεικνύει και την δέσμευση, την αφοσίωση των εθνικών υπηρεσιών να υποστηρίξουν την ε, χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο κύριος Μπράκε για την παρουσίαση των αστηριοτήτων σας. Κυρίες και κύριοι, είπα ότι ο κύριος Σάλμη θα χρειαστεί να φύγει ως τις 10 Οπότε πρότασή μου θα ήταν να κάνουμε τώρα τις ερωτήσεις, αν έχετε βεβαίως, στον κύριο Σάλμη. Αν έχετε λοιπόν, παρακαλώ, σηκώστε το χέρι σας ή τις καρτούλες που σας έχουμε δώσει. Ναι, παρακαλώ. Ο κύριος Ιγνάσιο Σάντσε, λέγομαι και έρχομαι από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή τον κύριο Σάμι. τρει φορέ επαναλάβατε και άρα θεωρώ ότι κρίνεται ότι είναι ένα βασικό στοιχείο για τη δουλειά τη ε, ε, ΙΝΣΕΝ ότι δεν συλλέγετε εσεί οι ίδιοι δεδομένα και ότι λειτουργείται σε θελούσια βάση και εισάγεται δεδομένα από τους εθνικούς, τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών. Λοιπόν, για μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, εγώ θα έκρινα λογικό να έχετε τα πετούμενα χέρια για να συλλέγετε και εσείς οι ίδιοι ε, δεδομένα. Θεωρείτε ότι είναι ευκταίο δεδομένου του επίπεδου ορίμανσης ε, των υπηρεσιών ε, πληροφοριών σε εθνικό επίπεδο, μήπως θα έπρεπε εσείς ε, σε ένα ρυθμισμένο πλαίσιο να έχετε τη δυνατότητα να συλλέγετε δεδομένα. Πιστεύετε ότι πρέπει να ανοίξει ένας τέτοιος διάβλος. Συγγνώμη, μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας γιατί δεν το ακούσαμε. Ιγνάθιο Σάντσες από την Ισπανική Βουλή. Κλοντ Συνάδελφοι, είναι εδώ οι κλητήρες και σας παρακαλώ να δίνετε το όνομά σας ε, στα καρτελάκια για να μην υπάρξει κάποια διακοινοβουλευτική σύγκρουση. Παρακαλώ να δίνετε το καρτελάκι με το όνομά σας ε, στους κλητήρες. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ. Καταρχάς θεωρώ δεδομένο και άκουσα ότι δεν ε, ε, διεξάγετε εσείς επιχειρήσεις. Εσείς τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγετε ε, τα αναφέρετε βεβαίως στην εκπρόσωπο αλλά και στις εθνικές υπηρεσίες και τι ακριβώς αξιολογείται την κατάσταση στις συγκεκριμένε ε, χώρες ε, όσον αφορά την ασφάλεια για, τους για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή για τις επιχειρήσεις που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα σύντομο ερώτημα. Συνεργάζεστε και με την Ευρωπόλ, την Ιντερπόλ και τις μυστικές υπηρεσίες τρίτων χωρών. Και μακροπρόθεσμα θα είχε νόημα να κάνετε δικές σας επιχειρήσεις ή θα ήταν καλύτερο ε, κάτι τέτοιο να συντονίζεται μέσω των εθνικών μυστικών υπηρεσιών. Ε, um, Και η κυρία Ίντφελτ έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υποθέτω ότι θα θέσουμε ερωτήματα μόνο προς τον εκπρόσωπο της Ίντσεν, έτσι δεν είναι. Ωραία. επανειλημμένα είχαμε, έχουμε συζητήσει αυτό το ζήτημα εδώ στο Κοινοβούλιο και ακόμη δεν έχω καταλάβει τι κάνει η Ίνσεν. Μας είπατε τι δεν κάνετε, αλλά εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τι όντως κάνετε. Ε, λέτε εμεί εμείς είμαστε σαν ε, θηρίδα, έρχονται υπηρεσίε πληροφοριών και μας βάζουν τις πληροφορίες μέσα και έρχονται κάποιοι άλλοι και τις παίρνουν». Ε, μα δεν είναι αξιόπιστο, δεν μπορούμε να σας πιστέψουμε διότι σε περίπτωση υπέρβαση αρμοδιοτήτων από τις υπηρεσίες πληροφοριών όπω διαπιστώθηκε όταν κατασκοπεύει το ένα κράτος μέλος το άλλο, κατασκοπεύουν ε, τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει στενή συνεργασία με τη CIA για έκνομε ε, δραστηριότητες. Και μετά την έκθεση της Γερουσίας ε, τον είπα για τις επιχειρήσεις CIA και τα βασανιστήρια, νομίζω Μα είπατε τότε, δεν έχουμε εμεί τρόπο να γνωρίζουμε ποια είναι η πηγή των πληροφοριών που λαμβάνουμε. Αυτό μας είχατε απαντήσει και τώρα έρχεστε σήμερα και μας λέτε «Άμα δεν χρειάζεται εποπτεία γιατί εμείς ε, διοικητικού χαρακτήρα δουλειά κάνουμε» όχι επιχειρησιακή, συγγνώμη, αλλά το ζητάω πάρα πολλά χρόνια να υπάρξει κατάλληλη εποπτεία και είναι καθήκον και του Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια όμως σε σχέση με το τι κάνει η Ινσεν, τι είδους πληροφορίες επεξεργάζεστε και ο Ισπανός συνάδελφος, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι Μπορεί ναι να μην συλλέγετε ατοπικά προσωπικά δεδομένα και σας πιστεύω δεν είναι αυτό, αλλά άλλο αυτό και άλλο το να μην επεξεργάζεστε ατομικά δεδομένα τα οποία προέρχονται από κάποιους άλλους. Ε, είστε πολύ καλός ε, ε, στο να επιλέγετε τη σωστή διατύπωση εγώ θα ήθελα μέσα στο πλαίσιο της συνθήκης, μέσα, στο πλαίσιο, ε, μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο να υπάρξει ε, εποπτεία. Σας ευχαριστούμε κυρία Ιντφέλτ, η κυρία Λόριστην. Ε, απηχώντας ε, το θέμα της Σόφη, τι ακριβώς κάνετε. Ποια είναι δική σας συνεισφορά. Συλλέγετε τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη αλλά την ανάλυση δεν την κάνετε για τα κράτη-μέλη όμως. Αν κατάλαβα καλά, την κάνετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα. Για την, για την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιες είναι οι βασικές απειλές γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για, μόνο για τα κράτη-μέλη. Και ποιο τμήμα, ποιο πόσο μεγάλο είναι το τμήμα της κύβερνο-ασφάλειας. Γιατί αυτό όπως ξέρουμε, είμαστε ε, σε μια περίοδο που υπάρχουν ε, πόλεμοι πληροφοριών, οπότε είναι μεγάλο το κομμάτι της ε, κυβερνοασφάλειας. Λοιπόν, σε αυτό το νέο περιβάλλον ποιες είναι οι απειλές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε κύριε Λόριστην. Ο κύριος Τούτσι τώρα από την Ιταλική Βουλή, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Σάμι. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για αυτό το σενάριο της υπηρεσία σε πληροφοριών και μπορείτε να σχολιάσετε τα θέματα κυβερνοασφάλειας και τρομοκρατίας αλλά ε, και δεν αγγίζω καν τις πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα για τον ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο πώς αντιλαμβάνεστε εσείς το ρόλο της INSEN δεν θα έπρεπε να αναθεωρηθεί ο ρόλος σε σχέση με τις τωρινές σας επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Στούτσερ. Κύριος ε, Σάλμη, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να προσπαθήσω να, καθα... να καλύψω όλες τις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, αν κατάλαβα καλά τη ρώτηση ο κύριος Σάντσες ε, για τα προσωπικά δεδομένα, και ε, απαντώ εν μέρη και στην κυρία Ιντβέλτ, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ούτε συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Και δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο για τις επιχειρήσεις μας και με ρωτήσατε, ε, λοιπόν τι κάνετε ε, ε αν δεν διεξάγετε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. 500 εκθέσεις συντάσσουμε όπως σας είπα και ε, τις μοιραζόμαστε ε, με την Ειδική Επιτροπή. Η ύπατη εκπρόσωπος ε, συσκέπτεται συχνά με την Ειδική Επιτροπή για να συζητά τις δραστηριότητές μας καθώς και τις εκθέσεις και νομίζω ότι λειτουργεί εύρυθμα το σύστημα προς το παρόν. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων. Ξέρω ότι ο Frontex και η Europol συγκεκριμένα λειτουργούν ε, μέσα σε ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο και για τις δραστηριότητες τους είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβούν ενδεχομένω σε μια τέτοια συλλογή προσωπικών δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μας αφορά αυτό. Ο κύριος Φως επίσης θα ε, κάνω μια, ένα, μια σχόλιο, γιατί όντω έπρεπε να το είχα αναφέρει. Ε, στέλνουμε τι εκθέσει μα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, μέσα από δύο διάβλους ε, στέλνουμε τις ε, εκθέσεις μέσα από τα υπέξε και από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Όλα τα ερευνητικά μας προϊόντα τα λαμβάνουν. Τώρα τα briefings που είναι πιο ειδικά έγγραφα τα επιφυλάσσουμε μόνο, τα, συγγνώμη, τα διαθέτουμε μόνο στην ΕΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και σε ε, άλλους ε, πελάτες ε, που έχουμε, που, τους οποίους διαφορούν άμεσα. Τώρα, γιατί μιλήσατε για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Δεν έχουμε καμία τέτοια αρμοδιότητα. Κάθε τέτοιο όργανο έχει δική του υπηρεσία. Είτε μιλάμε για την ασφάλεια του προσωπικού, για την ασφάλεια του κτηρίου, για την ασφάλεια των πληροφοριών ενίοτε λειτουργούμε συμβουλευτικά όταν υπάρχουν συγκεκριμένες απειλές και ε, αυτά ήθελα να σας πω για την κυβερνοασφάλεια. Ε, έχουμε επίσης εκπονήσει μελέτες ε, που απευθύναμε σε ευρωπαϊκούς φορείς. Εμείς προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε το θέμα, από πού προέρχεται η απειλή και πώς θα μπορούσαμε σε επιχειρησιακό επίπεδο να λειτουργήσουμε και προσπαθούμε να συμβουλέψουμε λοιπόν τα θεσμικά όργανα για θέματα κυβερνοασφάλειας. Για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες είναι πολύ περιορισμένη η συνεργασία, περιορίζεται ουσιαστικά στο εξή. Όπως σας έλεγα, βασιζόμαστε σε ε, συνεισφορές από τις ε, Εθνικές Υπηρεσίες Πληροφοριών και για να υπάρξει ανταλλαγή με ε, τρίτες χώρες πρέπει να ζητήσουμε συνένεση από αυτόν που εκπώνησε ε, την έκθεση ή μας έδωσε τα δεδομένα και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί τα κράτη-μέλη δεν επιθυμούν να έχουν τέτοια διμερή σχέση με τις τρίτες χώρες. Δεν είμαστε σε θέση να ε, ανταλλάξουμε εμείς πληροφορίες που έχουμε λάβει από τα κράτη-μέλη και το ίδιο ισχύει και για τις, ε, ε, τους υπόλοιπους ε, εθνικούς φορείς όπως ο εθνικός φορέας που βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης, εδώ στις Βρυξέλλες. Για την έννοια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι πολιτικό και νομικό το ζήτημα και ξεπερνά την αρμοδιότητά μου. Προς το παρόν όπως έχουν τα πράγματα είναι εθνική αρμοδιότητα οι υπηρεσίες πληροφοριών εάν κριθεί πρόσφορο να ακολουθήσουμε μια διαφορετική κατάσταση θα πρέπει να το αποφασίσει το Συμβούλιο και εγώ από ό,τι καταλαβαίνω θα, πρέ... θα επισύρει αυτό τροποποίηση της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Βραχυπρόθεσμα δεν προβλέπεται. Επίσης, ε, για τις δραστηριότητες και τις ανησυχίες μας. Όντως, κυρία Ιντβέλτε, ε, εδώ και καιρό συζητούμε τα ζητήματα αυτά και τώρα θα ήθελα να συζητήσουμε και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής ε, τη δυνατότητα να επισκεφτείτε το Ίντσεν και να δείτε από κοντά ακριβώς πώς διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας και τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια για να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα που, ή κάποιες ανησυχίε ε, που εξακολουθείτε να έχετε. Πρόεδρε, νομίζω, ελπίζω ως επιτοπλίστων να κάλυψα τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις. Ε, είστε ειδικό ε, και στη διαχείριση του χρόνου. Είναι 10 ακριβώς. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο David Bickford που είναι ο πρώην ε, νομικός διευθυντής ε, των υπηρεσιών, Βρετανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών MI5 και MI6. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα εδώ και είναι μεγάλη μου τιμή. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει βάλει τον πύχη αρκετά ψηλά όσον αφορά την ε, δέουσα ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγουν οι υπηρεσίε πληροφοριών πριν να αναλυθεί δράση επί τη βάση αυτών. Και αυτό γίνεται αποδεκτό από τι υπηρεσίε ε, πληροφοριών, γιατί αλλιώ αυτό θα αποτελούσε καταπάτηση των δικαιωμάτων των ε, ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων. Οπότε το αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε το ψηφιδωτό από τα στοιχεία τη ηλεκτρονική παρακολούθηση ε, και τι διάφορε άλλε αναφορέ. Αυτό γίνεται υποπίεση και πολλέ αυτό είναι δύσκολο, αλλά και ε, πάρα πολύ επικίνδυνο και ελέγχουμε και ξαναελέγχουμε και αναλύουμε πριν αναλάβουμε δράση επί τη βάση αυτών των πληροφοριών. Επίσης, ε, γι' αυτό το λόγο, ε, πριν ότι, ότι όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούμε να βρούμε για την ανάλυση μας, αυτό σημαίνει ότι θα πράγουμε και ανάλυση υψηλότερου επίπεδου. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική η ηλεκτρονική παρακολούθηση. Και θέλω να πω ότι το θέμα ε, είναι το που φτάνει αυτή η ηλεκτρονική παρακολούθηση και δεν μιλώ τώρα για την έγκριση αυτής ή για την εποπτεία της παρακολούθησης. Οπότε σήμερα έχουμε λοιπόν αυτούς τους ε, οργανισμούς και τις ομάδες που θέλουν να υπάρχει περιορισμός της παρακολούθησης αλλά ε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα μπορέσουμε να ανασχέσουμε τους τρομοκράτες. Θα πρέπει να έχουμε κάποιους μακρόπνες έρευνες και έχουμε επίσης και κάποιες αρνητικές πληροφορίες. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα στέλνει προσοχή μας στους στόχους. Επομένως να έχουμε όσο γίνεται λιγότερο κίνδυνο καταπάτηση των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων. Οπότε θα πρέπει τώρα να προβληματιστούμε για την λογική του επιχειρήματος το να περιοριστεί η ηλεκτρονική παρακολούθηση γιατί αυτό το οποίο απαιτείται από τις υπηρεσίες μας είναι να υπάρχει ανάλυση ψηλού επίπεδου. Άρα το ερώτημα παραμένει. Έχει κάποια σημασία, ή είναι χρήσιμη αυτή η ανάλυση. Η απάντηση είναι καταφατική, γιατί μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο φέτος έχουμε έναν ύποπτο για τρομοκρατία που συλλαμβάνεται κάθε μέρα. Πέρσι είχαμε 327 ε, που συλλάβαμε. 600 αναχώρησαν από το Ηνωμένο Βασίλειο για τη Συρία και δυστυχώς 300 ε, από αυτούς ήταν άγνωστοι στις αρχές. Έχουμε από το ίντερνετ χίλιες ιστοσελίδες τις οποίες κατεβάζουμε κάθε εβδομάδα. Οπότε θα πρέπει να καταπονήσουμε αυτό το οποίο ονομάζεται η δημιουργία ε, ενός πνεύματος ε, διαφθοράς ε, και παραπλάνησης των ανθρώπων. Και έτσι έχουμε κάποιους οι οποίοι περιθωριοποιούνται, γίνονται εγκληματίες, ε, αλλά και ευάλωτοι. Αυτά όλα θέλουμε να προστατεύσουμε και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την τρομοκρατία. Έχουμε αύξηση οργανωμένου εγκλήματο, έχουμε διακίνηση ανθρώπων, ε, δουλεμπόριο, εκπόρνευση ανηλίκων και όταν ήμουν ε, επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας των υπηρεσιών ε, πληροφοριών, ε, όλοι γνωρίζουν ότι είχα καλές σχέσεις με τις ομάδες προστασίας των δημοκρατικών ελευθεριών. Και είπαμε επομένως ότι θα πρέπει να δούμε πώς αυτές, αυτοί οι φορείς προστατεύουν τον κόσμο και όχι το να αποσπούν απλώς τα πρωτοσέλιδα. Θα πρέπει επομένως να υπάρχει κάποιο φορέα που να υποπτεύει τι υπηρεσίε πληροφοριών αλλά και τι ενέργειε που αναλαμβάνουν οι αρχέ επί τη βάση των πληροφοριών. Άρα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου ισορροπία και αυτό γίνεται επί τη βάση τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και έχουμε την υπόθεση Λάντερ κατά Σουηδία. Εκεί αναγνώστηκε από το δικαστήριο ε, το ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτή η ισορροπήση μεταξύ δικαιωμάτων και συλλογή πληροφοριών. Οπότε ζήτησε το δικαστήριο ότι θα πρέπει να υπάρχει νομοθεσία και έτσι να ε, καλυφθούν οι επιχειρήσεις και θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα μεταξύ του κινδύνου και του αποτελέσματος και επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια εποπτεία ε, του συνόλου πλέγματος αυτών των ε, υπηρεσιών. Αυτά τα είχα υποβάλει στα πλαίσια της εκδίκας της υπόθεσης Λεάντερ. Οπότε είπαμε ότι έτσι θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά του πέση πληροφοριών, αλλά και να περιορίζονται τα περιθώρια που υπάρχουν για κατάχρηση και καταπέραση δικαιωμάτων. Αυτό το οποίο απορρέει επίση, ε, αυτό που ακολούθησε τέλο πάντων την υπόθεση Λάντερ, έχουμε την υπόθεση Κλάσ. Κλάσ κατά Γερμανία στο 1978. Εκεί ε, κρίθηκε ότι η δικαστική εποπτεία ε, επί της παρακολούθησης είναι πιο ισόρροπη και είπανε ότι όταν οι εκτελεστικές αρχές ανακατεύονται με τα ατομικά δικαιώματα, τότε θα πρέπει να δει από την ενέργεια των αρχών από δικαστικό έλεγχο. Γιατί αυτό είναι καλύτερη εγγύηση ανεξαρτησίας, αμεροληψία και κάποιας ε, σωστής ε, διαδικασίας. Επομένως το πρόβλημα είναι ότι είχαμε την μαζική ε, εξέλιξη του ίντερνετ και σιγά σιγά Είχαμε όμως και την ανάπτυξη της κρυπτογράφησης και είχαμε αυτό που ονομάζουμε το σκοτεινό δίκτυο όπου χρησιμοποιείται από τους εγκληματίες και τους ε, τρομοκράτες και παρακάμπτουν τις αρχές ε, και επιτίθενται στην κοινωνία και στις ε, αξίες μας. Οπότε αυτό θα πρέπει να γίνει, να δούμε πώς θα μπορούμε να ασκήσουμε την, την παρακολούθηση για να προστατεύσουμε την κοινωνία και γι' αυτό και ε, αρχίσαμε να βλέπουμε τι γίνεται με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Επομένως τώρα έχουμε παρακολούθηση στα email, ε, στα website, στα κοινωνικά δίκτυα, ε, στην τηλεφωνία μέσω ίντερνετ, στα κινητά, παντού και επομένως τώρα ξεχάσετε ότι ξέρετε στο παρελθόν όσον αυτές τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις είχαμε, τώρα έχουμε το Communications Data Plus και ε, έχουμε τώρα κάποιον που μπορεί ε, να στείλει 100 ε, mail, να κοιτάξει ή να ανεβάσει 50 σελίδες στο ίντερνετ και 20 μηνύματα τηλεφωνικά. Αυτό το ονομάζουμε meta data. Και με, την εποπτεία τώρα έχουμε λοιπόν αυτή την αλυσίδα παρακολούθησης όταν κάποιος είναι ύποπτος. Και έτσι αυτό μας δείχνει και με ποιους σχετίζεται αυτός που παρακολουθούμε. Και γι' αυτό χρειάζεται ηλεκτρονική εποπτεία. Το θέμα λοιπόν ποιος θα δώσει την έγκριση για να γίνει αυτή η ηλεκτρονική παρακολούθηση και ποιος θα την εποπτεύσει. Ε, κάποιοι λένε ότι θα πρέπει το communication data plus να περιοριστεί και ότι θα πρέπει ε, η εποπτεία να είναι ακόμη πιο αυστηρή από ό,τι είπε το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων. Ε, ακόμα και όταν έχουμε κάποιο είδου διαμεσολαβητή επόπτη τον Αμίκου Σκούρια σύμφωνα με την Σύνδικη της Βενετίας οπότε χρειάζεται τώρα ε, ο, κάθε παρακολούθηση να περνάει από κοινοβουλευτικό έλεγχο. Στη ΔΕ Γερμανία έχουμε την, το, το νόμο G10 για το τι παρακολούθηση επιτρέπεται. Οπότε στην Γερμανία ε, μόνο οι ειδικοί δικαστές του, της αρχής εποπτείας των υπηρεσιών ε, παρακολούθησης που να δώσουν την άδεια. Οπότε αυτό γίνεται μόνο όταν υπάρχει κάποιο είδους ε, εύλογη ε, υποψία και βάσιμη εύλογη υποψία για κάποιον. οπότε έτσι παντού σε όλο τον κόσμο οι αρχές οι υπηρεσίε πληροφοριών καταπολεμούν την τρομοκρατία. Βεβαίως μιλάμε για ένα φαινόμενο διασυνοριακό ε, αυτό θα έλεγε ο χοντρός και ο λιγνός ότι αυτό είναι ένα υπέροχο χάος. Για να γυρίσουμε τώρα στην ε, απόφαση Λεάντερ. Όλα όσα είπε η υπόθεση Λεάντερ, όλα όσα έκριναν τότε οι δικαστές δεν ε, επηρεάζονται από την πρόοδο της τεχνολογίας. Γιατί έχουμε τώρα κάποιες περίπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης. Και όσο πιο περίπλοκες είναι αυτές όμως, τόσο πιο πολύ χάνεται χρόνος και ο χρόνος είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για την κατολέμηση της τρομοκρατίας. Οπότε έχουμε τώρα το θέμα της αναθεώρησης, της ε, τροποποίησης αυτών των ε, νόμων ή να έχουμε κάποιου νέε νέες υπηρεσίες πληροφοριών που να είναι διεθνείς ε, και να δούμε πώς μπορούμε αυτά να τα συμβιβάσουμε με την απόφαση Λεάντερ. Επομένω, είπαμε ότι τώρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουν δουλειά του υπηρεσίε πληροφοριών, αλλά θα πρέπει το εθνικό δίκαιο να αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι κάλυψη με πληροφόρηση ε, και παρακολούθηση ηλεκτρονική. Και επίσης χρειάζεται υποστήριξη από τα κοινοβούλια ή κάποια ανώτερη αρχή υποπτίας, ούτως ώστε να μην υπάρχουν καταχρήσεις και καταπατήσεις δικαιωμάτων. Επίσης έχουμε την απόφαση κλάση. Εκεί λέμε ότι έχουμε αυτό που ονομάζεται call face supervision στα αγγλικά. Δηλαδή είναι κάποιο είδους πρώτερη έγκριση. Και αυτό θα πρέπει να γίνει από τις δικαστικές αρχές και θα πρέπει ε, όμω να δούμε κατά πόσο να πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προβλήματα τη εκλογική εξουσία ή διπλωματικά προβλήματα. Αρνητική απάντηση. Οπότε θα πρέπει ε, ε, να θεωρηθεί ότι αν αυτά ελαμβάνονταν υπόψη θα είχαμε, κάτι, θα είχαμε παραλογισμό διότι έλεγε η, ε, η Βρετανική Επιτροπή Εποπτείας ότι οι δικαστές δεν είναι υπόλογοι για την εποπτεία και το Κοινοβούλιο ή κάποια άλλη ανεξάρτητη αρχή εποπτείας ε, έχει τελικά αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαδικασία διοδότησης. Επίσης, η Βρετανική Υπηρεσία Εποπτείας θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μια εκτελεστική αρχή που να ασκεί την ηλεκτρονική εποπτεία. Οπότε, τώρα μπορεί να έχουμε ε, παρακολούθηση χωρίς να υπάρχει αυτή η δικαστική άδεια. Γιατί είμαστε ως αρχές πληροφοριών υποπίεση για να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια του κόσμου. Επομένως θα πρέπει σε μερίσια βάση να λαμβάνονται οι αποφάσεις και η κρυφή παρακολούθηση έχει ως σκοπό ε, μοναδικό στο να καταπολεμήσει τρομοκράτες και οργανωμένο έγκλημα. Επίσης, όποτε υπάρχει συλλογή πληροφοριών από άλλα μέσα, αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ ε, ε, σημαντικό, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα στοιχεία αυτά και το θέμα είναι μέχρι πού μπορεί να διαβιβαστούν, μέχρι πού μπορεί να φτάσουν. Υπάρχει πίεση επομένως και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον η εκτελεστική αρχή είτε στην αρχή, στο τέλος της διαδρομής μπορεί να θεωρείται αξιόπιστη η αν είναι ανεπιθύμητη. Οπότε θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει το πώς γίνεται αυτή η εξορρόπηση των δικαιωμάτων σε σχέση με την απόφαση κλάσ. Η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θεωρεί ότι η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία της δημοκρατίας. Τώρα, η εκ των υστέρων εποπτεία δεν μπορεί να καλύψει όλες τις φάσεις της παρακολούθησης. Και ο δικαστής ε, Μπέρτον, που ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας της Επιτροπής Εποπτείας, είπε ότι θα πρέπει ε, να είμαστε βέβαιοι ότι όλα, ε, ο κάθε εποπτεία γίνεται υπό έλεγχο. Όμως, επειδή έχω δουλέψει πληροφοριών, μπορώ αυτό να το σεβαστώ. Το θέμα είναι ότι δεν είναι στεγανή ούτε αυτή η εκ των υστέρων εποπτεία. Επομένως, τώρα, ε, έχουμε προβλήματα από το Communications Data Plus, το Bulk Personal Data και αυτά οφείλονται στο πόσο γρήγορα ε, εξελίσσεται η ηλεκτρονική επικοινωνία. Οπότε χρειάζεται ε, και από τεχνολογικής πλευράς να ε, καλύψουν αυτή την πρόοδο με την κατάλληλη έγκριση. Και επίσης να υπάρχει μια ταχύτερη μέθοδος δικαστικής αδειοδότησης και έγκρισης. Και αυτό είναι θέμα τεχνολογικό. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς είναι οι δικαστές να εμπλακούν στις καθημερινές ενέργειες των υπηρεσιών πληροφορίας και να δίνουν επιτόπου, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή, την άδεια για παρακολούθηση και για αυτές τις ώρες τις, ε, ε, μυστικές ε, επιχειρήσεις. Και θα πρέπει επίσης αυτοί οι δικαστές να έχουν κάποιους συμβούλους ενεξάρτητους για να μπορούν να αποφασίσουν επί τη βάση των πιο πρόσφατων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Οπότε, έτσι, θα ήταν καλυμμένη η εκτελεστική εξουσία θα ήταν καλυμμένο το, το κοινό, ο κόσμος και οι φορείς των ανθρωπίνων, των δημοκρατικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα συμμορφωνόμασταν με τις αποφάσεις Λάντερ και, και Κλάς. Όμως γίνεται αυτό κάθε μέρα γιατί ε, μπαίνουν σε πειρασμό τα δικαστήρια να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο καταπάτηση των δικαιωμάτων και σε πολλές ε, περιπτώσεις έχουμε δικαστές υπηρεσίας πληροφοριών που εμπλέκονται σε επιχειρήσεις και ξέρουν τους στόχους και στενολογικές παραμέτρους. Έχουν εμπειρία δικαστές στο να σταθμίσουν ε, τις ενδείξεις και ε, στην σταδιοδρομία τους μπορούν να εξισορροπήσουν τα δικαιώματα από τη μια μεριά του κράτους και από την άλλη μεριά του ατόμου. Άρα θα πρέπει να δούμε κατά πόσον μπορεί να υπάρχει σε κάποια φάση ε, έρευνα από κάποιο ανώτερο φορέα ε, και από την άλλη μεριά να δούμε ποιο είναι πιο χρήσιμο. Δεν υπάρχει αυτός ο εξάρτητος φορέας ή ένας προσχετικός δικαστής που να δράει και επιτόπου. Και τελευταία φορά ε, συμφώνησα με τον Γάλλο συνάδελφο όσον αφορά το σύστημα που είχαμε προτείνει και από τότε όμως βλέπουμε ότι η γαλλική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια διαδικασία θέσπισης νόμων που καταργεί το προηγούμενο σύστημα και, και η ηλεκτρική εξουσία έχει αναλάβει στην ε, Γαλλία την ε, αδειοδότηση για ηλεκτρονική παρακολούθηση. Άρα η Γαλλία είναι στην εγκατάσταση με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε η νέα ε, νομοθεσία όπως ε, είπε ε, κάποιος διάσημος Γάλλος δικαστής στερείται κάλυψης από την νομολογία και από την πρακτική των δικαστηρίων. Οπότε βλέπουμε ότι είναι μεγάλη η πίεση στην εκτελεστική εξουσία, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και δύσκολο να διαχειριστεί η εκτελεστική εξουσία. Οπότε θα πρέπει οι υπηρεσίες να μπορούν να ενεργήσουν και θα πρέπει να μπορούν να υπάγονται σε κάποια δικαστική εξουσία. Να υπάρχει βοήθεια επίσης από εμπειρογνώμονες, τεχνοκράτες και από τα κοινοβούλια. Κύριε Μπίκφορ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε ε, ναι. Πολύ ενδιαφέροντος είπατε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν κάποιες ε, ερωτήσεις. Α, κύριος Βόητο. Εθνικός βουλευτής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσε οι απόψει που μας αναφέρατε εδώ. Ιδιαίτερα όσον αφορά ε, τα, ε, τους διάβλους που δεν είναι δημόσια προσβάσιμοι και είμαι σίγουρος ότι ε, αναφέρεστε και στη Γερμανία όπου εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης πολιτών και επιχειρήσεων και το ερώτημα μου είναι πού τελικά είναι ο έλεγχος γιατί εμείς ως Γερμανοί βουλευτές δεν έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε έλεγχο σε εσάς. Ε, Εσείς λογοδοτείτε δηλαδή στους, ε, στις Βρετανικές αρχές ή τελικά οι δραστηριότητες σας εμπίπτουν σε αυτήν την ιδιαίτερη κατηγορία της, ε, που δεν είναι δημόσια προσβάσιμες και δεν μπορούν να ελεγχθούν από δημόσιους φορείς. Ε, επόμενη ερώτηση από την κυρία Ιντφελτ. Πρόεδρε. Έχω πρώτα πρώτα προς εσάς κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα πρώτα όμως, μιλώντας γενικά, άκουσα το πάνελ. Ανησυχώ, γιατί θα έπρεπε να μιλούμε για την εποπτεία. Αλλά μέχρι τώρα το μόνο που ακούμε είναι ότι είναι άχρηστη η εποπτεία και σε μερικές περιπτώσεις μας λένε ότι είναι επικίνδυνη η εποπτεία. Μα με, νομίζω ότι κάπως οι υπηρεσίε πληροφοριών είναι σαν τις τράπεζες. Ότι δεν θέλουν ούτε μπορούν να διδαχθούν από όλα τα έχουν γίνει, τα διαβόντα μου για τα τελευταία χρόνια. Τι είναι, είναι τίποτα καουμπόιδες. Επίσης με σοκάρισε η εισήγηση της κυρίας Αμπολτίνα. Μα από ό,τι φαίνεται δεν έχετε ιδέα από το τι θα πει δημοκρατική υποπτία, ατομικά δικαιώματα. Οι υπηρεσίες είναι στην υπηρεσία του λαού. Δεν ισχύει το αντίστροφο. Γι' αυτό μιλάμε για δημοκρατική υποπτία. Ε, αυτό είναι που μας κάνει να διαφέρουμε από μια δικτατορία. Και μας είπατε ότι όλα είναι πάνω κάτω. Και τι γίνεται όσον αφορά ε, την κυβερνοεπίθεση στην Belgacom. Τι γίνεται με την έρευνα τη σχετική. Επίσης τι γίνεται με την έρευνα που αφορά τα μικρόφωνα που είχαν στήσει εδώ στο κτίριο του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες πριν από 10 χρόνια και ακόμα δεν ξέρουμε τι απέγινε η έρευνα. Επίσης για πέστε μας ισχύει ότι η εταιρεία που ασχολήθηκε με την κυβερνοεπίθεση στην Περγακόμ, η Ολλανδική εταιρεία Fox, ότι τους είπαν, επειδή ανακάλυψαν κάποια πράγματα, τους είπαν να κάνουν πίσω και ότι οι βελικές αρχές δεν θέλουν να στεναχωρούν τους Αμερικανούς και για αυτό και όλα αυτά τα κουκουλώσανε. Επίσης, είναι μια ερώτηση προς όλους σας. Μα πώς να να μας λέτε ότι δεν χρειάζεται η υποπτία ή ότι ό,τι ισχύει σήμερα είναι επαρκέσμα. Ξέρουμε τι έγινε με την Belgacom, τι έγινε με τις παραδόσεις της CIA κλπ. λοιπά Και μέχρι σήμερα ούτε μία ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν έχει στριμωχτεί να δώσει λόγο για ό,τι έκανε. Ενώ είχαν εμπλακεί όλα τα κράτη-μέλη και γνωρίζουν. τι γίνεται με τη συνεργασία των Γερμανών με την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί... Συνέχεια, τι ακούμε. Ακούμε για υπέρβαση εξουσία και κατάξη εξουσία από τι υπηρεσίε πληροφοριών. Άρα, τι είδου επιχειρήματα είναι αυτά που μα έχετε εκθέσει, ότι η εποπτεία σα εμποδίζει στι επιχειρήσει σα. Μα ήρθε η ώρα να υπάρξει κάποιο είδου αυθεντική εποπτεία. Και ο κ. Βόικτ έχει δίκιο ότι το πρόβλημα δεν είναι το τι γίνεται με την εποπτεία σε εθνικό επίπεδο. Είναι ακριβώς το θέμα το πώς διασυνοριακά συνεργάζονται οι υπηρεσίες πληροφοριών και αυτή η συνεργασία δεν είναι υπόκειται σε κανενός είδους εποπτεία. Μα εσείς υποτίθετε ότι προστατεύετε την ελευθερία και τη δημοκρατία. Είμαι πάρα πολύ ε, ανήσυχη και προβληματισμένη. Ευχαριστώ κύριε Νετβέλ, ο Θα λάβετε την απάντησή σα σε λίγο. Όμω, είχαμε τον κύριο Χάνς Κρίστιαν από τη Γερμανία, ε, επίσης ε, έτσι να μιλήσει. Είμαι ε, βουλευτής του Γερμανικού Κοινοβουλίου, το όνομά μου είναι και είμαι και μέλος της Επιτροπής ε, για ελέγχου των ε, μυστικών υπηρεσιών και της Επιτροπής, της Ειδικής Επιτροπής που έχει συστηθεί για την υπόθεση NSA. Και ο κύριος Μπάκη αλλά και ο κύριος Μπίκφορτ ανέφεραν ε, ότι ε, είναι σημαντική, σημαντικός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ε, αναφέρθηκε από τον κύριο Μπράκη ότι και οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει να παραδίδονται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές όταν διεξάγεται ένας τέτοιος έλεγχος. Τι γίνεται όμως στην πράξη. Στην πράξη όταν η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση αποστέλει ή πρέπει να δώσει πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα στην ε, Εξεταστική Επιτροπή, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου απειλεί να διακόψει τις ε, σχέσεις μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών αν η γερμανική κυβέρνηση παραδώσει εμπιστευτικές πληροφορίες ή έγγραφα στην Εξεταστική Επιτροπή της ε, Γερμανικής Βουλής. Αυτό γίνεται στην πράξη. Όλα τα άλλα ε, είναι θεωρία. Και δεν καταλαβαίνω γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και άλλα εθνικά κοινοβούλια δεν ασχολούνται περισσότερο με το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία υπάρχει η αιτιολογημένη υποψία ότι ε, η NSA κατά τις διαδικασίες ε, της εργασίας παρακολούθησης της στην Ευρώπη με τη βοήθεια των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών παρακολούθησε Γάλλους πολιτικούς ε, εργασίες ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αλλά και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Ενώ αποδεικνύεται μέσα από το θέμα αυτό πόσο σημαντική είναι η συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών της Ευρώπης και πόσο σημαντικό είναι να βρεθούν τρόποι ώστε οι επιτροπές ελέγχου των εθνικών κοινοβουλίων μπορέσουν να συνεργαστούν περισσότερο μεταξύ τους προκειμένου να ε, ασχοληθούν με ζητήματα όπως ε, αυτά που ε, ανέκυψαν με την NSA στη Γερμανία. Ευχαριστώ κύριε Στρόμπελε. Ο κύριος Μωράης. το ερώτημά μου απευθύνεται στον κύριο Μπίκφορντ και τον κοινοβουλευτή κοινοβουλευτικό έλεγχο, την κοινοβουλευτική εποπτεία. Αλλά ε, υπό το φως και αυτών που ακούστηκαν από τους συναδέλφους, θέλω να πω το εξής. Η έρευνα που διεξήγαγε το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ε, αρμοδιότητα. Εμείς αυτό που κάναμε και ερευνήσαμε ήταν τι γίνεται όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στα κράτη-μέλη. Η κυρία Ινβέλτ ε, έδωσε ένα παράδειγμα για το Βέλγιο συγκεκριμένα. Εμείς όμως καλούμε να ενισχυθεί η εποπτεία και αξιοποιούμε όλη την πολιτική επιρροή που έχουμε για να μεταρρυθμιστεί το αναχρονιστικό πλαίσιο που υπάρχει σε μια σειρά κράτη-μέλη. Αυτό κάνουμε και δεν ε, μπορούμε ωστόσο να υποκριθούμε ότι έχουμε νομικές εξουσίες που δεν έχουμε. Κύριε Μπίκφορντ, ε, ένα ερώτημα σας. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας από ό,τι κατάλαβα, δεν ξέρω αν το είπε και η Σόφη, ε, ήταν ότι αυτό που κάνατε ε, ήταν να παρουσιάσετε ε, λεπτομερώς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, την κοινοβουλευτική εποπτεία. Στη Γαλλία υιοθετείται μία, ένα καθεστώς που ισχύει και στην, στη Βρετανία. Υπάρχει ένα εξαιρετικά περίπλοκο καθεστώς, ε, ένα σύστημα μαζικής συλλογής πληροφοριών ε, μέσα από το DCHQ ε, ενώ ταυτόχρονα το, το καθεστώς κοινοβουλευτικής εποπτείας είναι αναχρονιστικό και δεν έχει μεταρρυθμιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με άλλα λόγια το κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση, ακόμη και αν έχει την πρόθεση ή τη θέληση, δεν μπορεί να ε, ανταποκριθεί σε αυτό το τεράστιο ε, έργο που έχει μπροστά του να επιτελέσει. και το ερώτημά μου είναι το εξής το δικαστικό μοντέλο που προτείνετε, που προτείνετε μάλλον εσείς είστε υπέρ αυτού γιατί σε κάποιες περιπτώσεις ούτε οι δικαστές δεν θα έχουν τη δυνατότητα δεδομένου του τεχνικού και του τεχνολογικού χαρακτήρα των γνώσεων που χρειάζονται για να αντιμετωπίζει και να εξετάζει κανείς τέτοιου είδους ζητήματα. Ε, Καταλαβαίνετε τι λέω, δεν θα μπορούν οι δικαστές οι ίδιοι να ανταποκρίνονται στις, ε, στις ε, υποθέσεις που τους ανατίθενται. Λόγω της περιπλοκότητάς τους. Οπότε τι είδου κοινοβουλευτική υποπτία θα πρέπει να προτείνουμε εμείς. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμείς θέλουμε να δώσουμε συνέχεια και στην έκθεσή μας. Διότι γνωρίζουμε ε, ότι υπάρχει ε, δημοκρατικό έλλειμμα, ε, έλλειμμα όσον αφορά τη, την τεχνική πλευρά του ζητήματος. Οπότε το, το ερώτημά μου είναι ποιο, ποιο θεωρείτε εσείς ότι θα ήταν το καλύτερο μοντέλο που θα πρέπει να προτείνουμε. Γιατί ανησυχώ για αυτό που συμβαίνει στην, στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, διότι υιοθετείται εκεί ένα βρετανικό σύστημα, το οποίο όμως ε, από προβλήματα. Ευχαριστούμε κύριε Μωρές. Θα ακούσουμε πρώτα όλες τις ερωτήσεις και μετά τον κύριο Μπίκφορντ, Η κυρία Καλυμέντε από τη Ρουμανία. Yes, please. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Καλυμέντε. Αξιότιμοι βουλευτές. θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η σημερινή μας διάσκεψη, διότι πέρα από τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, το διακύβευμα είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η σημερινή διάσκεψη. Συζητούμε όλοι για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των υπηρεσιών πληροφοριών Ακριβώς επειδή θα πρέπει να υπάρχει ε, μη στρατιωτικός έλεγχος των υπηρεσιών πληροφοριών. Πρόκειται για μια πάγια ανησυχία της ε, Ρουμανικής Βουλής. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας η μόνη κοινοβουλευτική συνέλευση της Δυτικής Ευρώπης ε, που είχε αρμοδέτα για τέτοια ζήτημα δεν υφίσταται πια. Δεν υπάρχει πλέον συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών και νομίζω ότι παρατηρούμε όλοι τις ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί σε αυτό το τομέα με τις νέες προκλήσεις, τα μεταναστευτικά ρεύματα από τη Βόρεια Αφρική, με τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Ευρώπη, την επίθεση της ε, Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και ούτω καθεξής. Μας απασχολούν επίσης ε, θέματα που σχετίζονται και με την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όλοι αναφέρονται σε προβλήματα, καλό θα ήταν όμως να ακούσουμε επιτέλους και κάποιες απαντήσεις. Καλά όλα αυτά που λέμε, όμως εν τέλει είναι ένας ε, σημαντικός σύμμαχός μας ε, στο ΝΑΤΟ ή Σίγουρα όλοι φοβόμαστε την τρομοκρατία, την παράνομη μετανάστευση, όλες τις ε, σύγχρονες απειλές, όμως γιατί δεν φοβόμαστε ένα ε, κράτος που είναι επιθετικό και επιτέθηκε ήδη σε μια χώρα. Μιλώ φυσικά για τη Ρωσία. δεν πρόκειται εδώ για ηλεκτρονική κυβερνοεπίθεση, όμως ε, γίνεται ένας πόλεμος στο διαδίκτυο στη διάσκεψη του ε, Βίλνιους. Ανατέθηκε στην Ρουμανία να αναλάβει το συντονισμό της ε, άμυνας μέσω ηλεκτρονικών μέσων και θα ήθελα να ρωτήσω μετά από αυτήν την μαζική επίθεση της Ρωσίας μέσα από ηλεκτρονικά μέσα, ποια απάντηση τελικά δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπιστώνω ότι δεν ασχολούνται πολύ με αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις με της Ρωσίας. Πρόσφατα με την ιδιότητα του βουλευτή μετέβη στην Ουκρανία και μπορώ να σας ενημερώσω ήδη ότι δεν θα σταματήσουν οι Ρώσοι. Ε, ετοιμάζουν ήδη την επόμενη επίθεση για τη Μάριοπολ και χρησιμοποιούν ε, όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, μεταξύ των οποίων και οι κυβερνοεπιθέσεις. Κάθε κράτος μέλος έχει καθήκον να αντιδράσει, όμως πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και μια συλλογική απάντηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λέει κυρία Κρίσπεκ. Ευχαριστώ τον Κλοντ Μορέσε που διοργάνωσε τη σημερινή συνάντηση είναι ευπρόσδεκτη όχι μόνο στα πλαίσια της ε, πάγιας διαθεσμικής συνεργασίας με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία διότι είναι εξαιρετικά επίκαιρα τα ζητήματα και μεγάλες οι απειλές που αντιμετωπίζουμε, οι τρομοκρατικές επιθέσεις ε, που ε, δυστυχώς αποσχολούν την επικαιρότητα. Βλέπουμε ότι συντρέχει συντρέχουν πολλοί λόγοι για να ε, ασχοληθούμε με αυτά τα οριακά θα έλεγα μέσα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες ε, πληροφοριών για να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές. Στις αρχές ε, του Μαΐου πέρασε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή για την υπηρεσία πληροφοριών μέσα από μια ευτυχημένη διαδικασία και δεν θα το σχολιάσω αυτό, το θέμα δηλαδή της διαδικασίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν συνάδελφοι από το, την, Εθνική, ε, την Γαλλική Εθνοβουλή, Εθνοσυνέλευση και μπορούν να σχολιάσουν αυτό το νομοσχέδιο που παρουσιάζει ο πρόεδρος Ολάντε και ε, το υπέβαλε στο Συμβούλιο Επικρατείας ε, για να εξεταστεί η συνταγματικότητα αυτού του νομοσχεδίου. Συζητείται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και κατά πάσα πιθανότητα θα υιοθετηθεί και δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Κάποια από αυτά αναφέρθηκαν και προσθέτω το εξής ε, υπερβολική επέκταση των αρμοδιοτήτων του αρχηγού της κυβέρνησης απουσία απριόρι ε, ενός δικαστικού ή ακόμη και διοικητικού συστήματος ελέγχου ε, μέσα από ένα σύστημα μαζικής ε, υποκλοπής και παρακολούθησης δεδομένων από Πλευρά των πολιτών για περαιτέρω ανάλυση. Έχουμε και το άρθρο 66 του Γαλλικού Συντάγματο που προβλέπει ότι οι δικαστικές αρχές είναι οι θεματοφύλακε των βασικών ελευθεριών και των προσωπικών ελευθεριών. Όμως ε, δεν υπάρχει εισαγγελέα, δεν έχει ρόλο εισαγγελέα μέσα σε αυτό το σύστημα υπερβολικού, υπερβολικών αρμοδιοτήτων ε, για τον αρχικό κυβέρνηση ω προς τι Υπηρεσίε πληροφοριών. Και μην ξεχνάμε ότι ε, καμία τέτοια διάταξη αντιβαίνει και στην ομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, αντιβαίνει και στις συνθήκες. Για να μην μακρηγορώ, αυτή η απουσία δικαστικού ελέγχου ε, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τη γνώμη σας, σε πώς τοποθετήσετε σε σχέση με αυτό, πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε ε, στα πολλαπλά αιτήματα ελέγχου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμη και αν κατοχυρωθεί ο δικαστικό έλεγχο, δεν υπάρχουν αρκετοί δικαστέ, δεν υπάρχουν ε, τα απαιτούμενα μέσα για να ανταποκριθούμε στον αυξανόμενο αριθμό ετοιμάτων. Σα ευχαριστούμε, ο κύριο ε, Γκαλασεύσκη από την Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθώ τη συζήτηση και να σας πω ποιες είναι οι σκέψεις μου. Πρώτα πρώτα. Επιβάλλεται να υπάρχει υποπτία. Χρειάζεται έλεγχος επί των υπηρεσιών πληροφοριών. Όμως, από την άλλη μεριά, θέλουμε αυτές οι υπηρεσίες να γίνονται πιο αποτελεσματικές. Μας έχει διδάξει η ιστορία μας τους Πολωνούς ότι ε, όχι μόνο εμείς, αλλά και άλλους λαούς το ότι πάρα πολύ εύκολα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τους πολιτικούς στο παρελθόν. Είχαμε ένα σωρό κατάσκοπους που ε, ασχολούνται με την πολιτική στην κομμουνιστική Πολωνία, οπότε βλέπουμε πώς εξισορροπούνται τα πράγματα τώρα βέβαια αλλάζουν κάπως τα πράγματα, αλλάζει το τοπίο. Άρα, θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη πρόσβαση στην πληροφορία. Χωρίς πληροφορία βέβαια δεν μπορεί να υπάρχει εποπτεία. Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο κάνει η Νορβηγία που υπάρχει κοινοβουλευτική επιτροπή, ε, εκλέγεται από το κοινοβούλιο, αλλά τα μέλη της ε, επιτροπής αυτής είναι κάποιοι ανεξάρτητοι, είναι κάποιοι που δεν ανήκουν σε κόμματα. Να ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Και εγώ πολιτικό είμαι, αλλά πιστεύω ότι οι πολιτικοί δεν θα πρέπει να έχουν τόσο πολύ λιμένα τα χέρια τους ε, στο θέμα της, ε, της, της εποπτείας. Έχουν άλλα πράγματα να κάνουν. Έχασε το και ο πρώτο και τώρα έχουμε άλλου δύο οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο, ήδη τον έχουν ζητήσει και θα θέλουν να δευτερολογήσουν. Οπότε παρακαλώ να είναι σύντομοι. Στούτσια. Το Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σημαντικό το θέμα. Μα γι' αυτό και έχουμε τόσες ε, παρεμβάσεις και ερωτήσεις. Θέλω να σας πω ότι χρειάζονται δύο τύποι εποπτείας και ελέγχου. Πρώτα πρώτα συγκεκριμένος έλεγχος από τους ε, δικαστές για κάποια ζητήματα που αφορούν τις ατομικές ελευθερίες. Οπότε χρειάζεται να γίνει τέτοια επιλογή για την άλλη μεριά. Έχουμε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, εκεί που είναι πιο πλήρε πιο εξαντλητικός ο έλεγχος. Επίσης τώρα το θέμα είναι το πώς ε, θα ενημερώνεται το κοινό για όλα αυτά, γιατί υπάρχει εδώ πέρα το θέμα του απορρίτου. Θα πρέπει να καταλάβει κανείς το ότι η δραστηριότητα των υπηρεσιών αυτών αφορά κάποια πολύ λεπτά ζητήματα, κάποια βρώμικα ζητήματα. Ε, πολλές φορές ε, σκέφτομαι ότι μόνη δυνατότητα να έχουμε μία έλεγχο από κοινοβούλιο είναι το να υπάρχει ε, έγκριση από το Κοινοβούλιο στον αυτό τον προϋπολογισμό αυτών των υπηρεσιών. Γιατί πού να έχουμε καθαρές απαντήσεις για το πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες. Ε, οπότε η Επιτροπή, το όργανο ελέγχου τέλος πάντων, ε, του ελέγχου επί των υπηρεσιών αυτών που ελέγχει και εκ των υστέρων εγκρίνει, θα μπορεί να πει μπλοκάρουμε την πρικοδότηση γιατί δεν είμαστε σίγουροι τι κάνετε, αν αυτά που κάνετε αντιστοιχούν στα συμφέροντα της χώρας ή ε, γιατί δεν θεωρούμε ότι όλα όσα κάνετε συνάδουν προς τη δημοκρατία. Τώρα όσον αφορά την πρικοδότηση για μένα ε, αυτό είναι το πιο λεπτό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το μελετήσουμε για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα, στα ερωτήματα τα σχετικά με τις παρεχόμενες εγκλήσεις. Ποια πέστε μας τη γνώμη σας. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βόητ τώρα θα δευτερολογήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος ε, Στρόμπελ επιβεβαίωσε πριν από λίγο ότι το Ενωμένο Βασίλειο ε, απειλεί να διακόψει τις επαφές με τη Γερμανία προκειμένου να παρεμποδίσει την παροχή πληροφοριών στις εξεταστικές επιτροπές ε, της Γερμανικής Βουλής. λόγω των ειδικών διατάξεων που ισχύουν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ε, πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν ε, Γερμανούς πολίτες και επιχειρήσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος ελέγχει, ποιος σας ελέγχει όσον αφορά την συλλογή των πληροφοριών εκατομμυρίων Γερμανών πολιτών. Ε, πρώτα απ' όλα, πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Μπίκφορτ. Θα ήθελα να απαντήσω, λέει ο κύριος Μπράκε, ε, ως πρόεδρος, σε κάποια ερωτήματα που τέθηκαν από την κυρία Ίνφελτ και θα σας ε, απαντήσω στα Ολλανδικά, για να είμαι όσο πιο ακριβή γίνεται. Λοιπόν, να ξεκινήσω και να πω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι σαφές ότι θα υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ της ε, πρακτικής ε, των ε, μυστικών υπηρεσιών και του δημοκρατικού ελέγχου. Αυτό είναι φυσιολογικό και για τα επιμέρους ερωτήματα που θέσατε. Νομίζω ότι τα ζητήματα που θέσατε συγκεκριμένα για τα μικρόφωνα που βρέθηκαν στο κτίριο γιους τους λήψης υπάρχει νομική έρευνα η οποία μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και το θέμα έχει τεθεί στο αρχείο. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να δοθεί συνέχεια σε αυτό. Όσον αφορά την έρευνα για την ακόμη εκκρεμεί ακόμη. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι και στα δύο ζητήματα που θίξατε ε, έχει υπάρξει έκθεση από την επιτροπή, τη μόνιμη επιτροπή I και στις δύο εκθέσεις υπάρχουν παρατηρήσεις που αφορούν τις δικές μας μυστικές υπηρεσίες και αναφέρεται ότι θα έπρεπε να είχαν αναλάβει πολύ πιο δραστήριο ρόλο. Και βεβαίω οι πληροφορίες αυτές θα διαβιβαστούν και στις ίδιες μυστικές πληροφορίες και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από αυτές. Και τέλος να πω ότι στο Βέλγιο έχουμε τη μόνιμη επιτροπή ΆΗ για τις μυστικές υπηρεσίες και για λόγους σύγκρισης μπορώ να σας πω ότι αυτές, αυτή η επιτροπή, η δική μας επιτροπή δηλαδή, ασκεί ε, εκτεταμένο έλεγχο και συγκριτικά και με αντίστοιχες επιτροπές από άλλες χώρες. Και παρακολουθούμε τις τεχνικές και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και τις ελέγχουμε. Υπάρχει ομολογώ, ένα πρόβλημα ή διάφορα προβλήματα. Αλλά η διάσκεψη μας σήμερα ε, έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης γιατί δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα επί μυστικών υπηρεσιών άλλων χωρών που δραστηριοποιούνται στη δική μας επικράτεια. Ε, και φαίνεται νομίζω ότι υπήρξε και άλλο ένα ερώτημα από τον κύριο Ζετικόφσκι αν το προφέρω σωστά θα του δώσω το λόγο σε λίγα δευτερόλεπτα αλλά θέλω να ε, επισημάνω ότι ο πρόεδρος του Επιτροπής, ο σήμερα, στη διάρκεια της ε, ημέρας, θα σας δώσει και μια έρευνα για το τι κάνουμε και πώς το κάνουμε. Λοιπόν, πρωτού δώσω το λόγο στον κύριο Μπίκφορτ, μια τελευταία, ε, τελευταία ερώτηση από τον κύριο Ζεντόφσκι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Πρώτα απ' όλα, να πω ότι ε, εργαζόμουν για το Υπουργείο Συντερικών της Τσεχίας και εκεί υπήρχε ένα αστείο ότι ένας πολιτικός που δεν βρίσκεται υπό, επιτήρηση είναι είτε άχρηστος είτε μη ενδιαφέρον. Αλλά πέρα από την πλάκα είναι πολύ σοβαρό το θέμα που συζητούμε σήμερα. Κατά τη γνώμη μου οι δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών ε, θα πρέπει να παρακολουθούνται και μάλιστα σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το επαγγελματικό επίπεδο. Κανένας δικαστής, κανένας πολιτικός δεν μπορεί να αξιολογήσει με ορθό τρόπο την ε, χρήση, για παράδειγμα, συγκεκριμένων τεχνικών μέσων στην ε, συλλογή πληροφοριών στην οποία προβαίνουν μυστικές ε, υπηρεσίες. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, όπου, για παράδειγμα, πρώην διευθυντές μυστικών υπηρεσιών θα μπορούσαν να συμμετέχουν ή θα μπορούσαν να συμμετέχουν κάποιοι με αδιαμφισβήτητα διαπιστευτήρια ε, στον τομέα αυτό. Ε, αυτό που είπε η Σόφη καταδεικνύει ότι εμείς ως πολιτικοί θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε να υπάρχει έλεγχος και εποπτεία των βασικών αρχών της δημοκρατίας. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που συζητούμε σήμερα και το ανέφεραν και πολλοί συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι το γεγονός ότι οι πολιτικοί δεν θέλουν να κάθονται και να ελέγχουν την κάθε απόφαση των μυστικών τους υπηρεσιών. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να διασφαλιστεί ότι οι μυστικές υπηρεσίες δεν ελέγχουν το που βρίσκεται ο καθένας ή δεν αξιοποιούνται στις συγκρούσεις μεταξύ πολιτικών. Αλλά έχω και μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ω σύνολο. Οι μυστικές υπηρεσίες των κρατών μελών εμπιστεύονται η μία την άλλη ή αντιμάχονται η μία την άλλη. Μήπως εξακολουθούμε να ζητούμε τον, ε, τον ε, εχθρό εντός. Αυτό μας ανησυχεί. Υπάρχουν 28 κράτη-μέλη που το καθένα τους έχει πράκτορες στα άλλα κράτη-μέλη ε, φαίνεται δηλαδή να υπάρχουν κάποια απομεινάρια του ψυχρού πολέμου σαν να έχει παγώσει ο χρόνος πριν από 25 χρόνια. Και ένα ακόμη ερώτημα τεχνικού χαρακτήρα. Κρυπτογραφημένες επικοινωνίες δεν έχουν ανεφερθεί καθόλου μέχρι τώρα, αλλά γνωρίζω ότι για τις μυστικές υπηρεσίες ε, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτό. Πώς δηλαδή μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ε, πληροφορίε για τρομοκρατικέ οργανώσει που είναι κρυπτογραφημένε και νομίζω ότι η εποπτεία σε αυτό το, σε αυτό το τομέα δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι πολιτικού χαρακτήρα, πρέπει να έχει τεχνικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι κάποια από τα ερωτήματα που θέσατε μπορούν να τα απαντήσει και ο επόμενος ομιλητής. Δεύτερον, θα ήθελα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Αμπολτίνα γιατί αναφέρθηκε και εκείνη από την ε, κυρία Ίντφελτ. Θέλω κυρία είναι, να σας πω ότι στην ομιλία μου αυτό το οποίο ήθελα είναι να σας πω ότι δεν χρειάζεται καν η εποπτεία, όταν αυτό, λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και άρα θα πρέπει εμείς που εποπτεύουμε τις υπηρεσίες να συνεργαστούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι υπηρεσίες πληροφοριών να συνεργάζονται μεταξύ τους. Παρεξηγήσατε αυτό το οποίο έλεγα. Αν επομένω δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο οι υπηρεσίε πληροφοριών, ε, τότε φυσικά και χρειάζεται να έχουμε εποπτείε. Αλλιώ θα έχουμε του ε, καταδότε, του πληροφοριοδότε που θα του εκθέσουν. Τι υπηρεσίε δηλαδή εννοώ. Οπότε θα πρέπει όλοι, όλοι να σέβονται τον νόμο. Όλε οι πλευρέ. Ευχαριστώ κυρία Μπολτίνα. Κύριε Μπέκφορντ, εσεί τελευταίο. Ευχαριστώ πρόεδρε. First thing 100% με όλους τους προβληματισμούς που εξετέθησαν και προσωπικά δεν πιστεύω ότι το επίπεδο εποπτείας ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υψηλού επίπεδου. Συμμορφώνεται η εποπτεία ε, με την απόφαση Γκάντερα αλλά όχι ε, με, με τα όσα έκρινε το δικαστήριο στην απόφαση Κλάς. Βέβαια, αυτό δεν πάει να πει ότι όλα τα κράτη που έχουν υποπτία δεν κάνουν ό,τι μπορούν για να ελέγξουν τις υπηρεσίες. Ξέρουμε τι προβλήματα ανακύπτουν όταν ε, είναι εκτός ελέγχου υπηρεσίες πληροφοριών. Άρα, θέλω να σας πω το εξής. executive authority. Η εκτελεστική εξουσία ας πούμε ο αρμόδιος υπουργός που εποπτεύει τις ε, επιχειρήσεις δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι ανεπιθύμητος ο έλεγχός του. Είναι αναξιόπιστος. Ε, δεν θα πρέπει αυτός ο έλεγχος να θεωρείται επομένω βάση και κάτι το αξιόπιστο. Τώρα παρακάτω. Έχουμε δύο επίπεδα. Ε, δύο θέματα που είπε ο Ιταλός συνάδελφος. Έχουμε το δικαστικό έλεγχο και από την μεριά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα, ποιες είναι οι δυσκολίες, ποια είναι τα προβλήματα όταν ανακατεύονται με τα δικαιώματα οι υπηρεσίες. Ότι αυτό γίνεται την ώρα που έχουμε τις επιχειρήσεις. Ή μάλλον καταπάτηση δικαιωμάτων μπορεί να έχουμε και πριν αρχίσουν οι επιχειρήσεις. Εάν η υπηρεσία θεωρεί ότι πρέπει να προβεί σε κάποιες ενέργειες, σε κάποια επιχείρηση που φύγει ατομικά δικαιώματα, τότε είναι αργά να υπάρξει εποπτεία. Μα ήδη έχει γίνει ενδεχομένω αυτή η επιχείρηση, γιατί ήδη έχουν αναμειχθεί υπηρεσίες με το άτομο, με το κάποιο φυσικό πρόσωπο. Μπορεί κανεί εκ των υστέρων να προσπαθήσει να καταστήλει, αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Αυτό που θέλουμε και προτείνουμε είναι η έγκριση να δίνεται πριν η υπηρεσία αναμειχθεί με το φυσικό πρόσωπο. Και αυτό μπορεί να γίνει με κάποιο είδου ηλεκτρονική εποπτεία. Πώ μπορεί να γίνει αυτό από το κοινοβούλιο, ε, δεν νομίζω. Πόσοι από εσά έχετε χρόνο κάθε μέρα να παρακολουθείτε, να ακούτε τι λένε στις υπηρεσίες που θα αναμειχθούν με κάποιο άτομο και τα δικαιώματά του. Άρα θα πρέπει να βρεθεί μια εναλλακτική λύση. Ποια είναι αυτή. Προτείναμε να το κάνουν αυτό πρώην πράκτορες των υπηρεσιών. Αυτό όμως πιστέψτε με δεν είναι η άριστη των λύσεων οι πράκτορες, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών πληροφορίων θέλουν να μας προστατεύσουν. Υπάρχουν τρόποι. Άρα θα πρέπει να υπάρχει, ας το πούμε, αυτοέλεγχος. Επομένως, ποιος άλλος υπάρχει που θα μπορούσε να βοηθήσει κάποια επιτροπή με νομικούς και πολιτικούς. Θα πρέπει όμως να συνέρχονται αυτοί, να συνδυάζουν καθημερινά. Πού όμως, μα οι πράκτορες πάνε παντού για να μπορούν να ε, παρουσιάσουν το τι κάνουν. Και τι θα πούνε στην Επιτροπή αυτή. Θα τους πούν ό,τι μπορούν. Και ποιος θα ε, αντιλέγει. Ποιος, ε, αυτός ο ειδικός επίτροπος Αμίκος Κούριε. Μα αυτόν θα τον ε, αντιμετωπίσουν οι αρχές των πληροφοριών θα το ανατρέψουν επιχειρήματα. Τότε τι απομένει. Απομένει, λέω, να υπάρχει κάτι όπως κάνουν οι δικαστές. Να είναι κάποιος δικαστικός. Το κάνουν αυτό οι Γάλλοι και δυστυχώς θέλουν τώρα να το καταργήσουν και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ανόητο. Αυτός λοιπόν ο ανακριτής ας πούμε, ο οποίος, ο οποίος θα εδρεύει μέσα στην υπηρεσία πληροφοριών, αυτός λοιπόν θα είναι εκεί και θα παρακολουθεί το σύνολο της διαδρομής μιας επιχείρησης. Και δεν είναι το θέμα μόνο η ηλεκτρονική παρακολούθηση, η εποπτεία. Έχουμε παρακολούθηση μέσα σε κτίρια, έχουμε πληροφορίες που έρχονται από έξω από την υπηρεσία και αυτό ο δικαστικός, αυτός ο ανακριτής παρακολουθεί. Και ακριβώς επειδή είναι εκεί, μέσα στην υπηρεσία, είναι η θέση να μπορέσει να κρίνει πότε και εάν Έχουμε καταπάτηση ατομικών δικαιωμάτων ή τέλο πάντων επικείμενη καταπάτηση ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί να έχει κάποιον ε, τεχνοκράτη να τον ε, συμβουλεύει, κάποιον εμπειρογνώμονα, δεν είναι δύσκολο. Άρα είναι εκεί επιτόπου. Τώρα, πέραν αυτού, θα πρέπει να υπάρχει κοινοβουλευτική εποπτεία ή κάποιο είδου αμερόληπτη αντικειμενική ή ανεξάρτητη εποπτεία. Οπότε όταν έρθει η ώρα να υπάρχει αυτό το σώμα, αυτό ο φορέα να κάνει κάποια έρευνα και να καλεί κάποιους από την υπηρεσία πληροφοριών για να τους ούτω επί να ανακρίνει για να του υποβάλει ερωτήσει και να καλύπτονται και τα θέματα τη προποδότηση του προπολογισμού. Γιατί ένα από τα θέματα με τι υπηρεσίε πληροφοριών είναι ότι έχουν περιορισμένο προπολογισμό. Δεν έχουν τα εκατομμύρια, τα δολάρια ή τι λίρε ή τα ευρώ στη διάθεσή του. Έχουν περιορισμένη προποδότηση. Εγώ έχω εξετάσει πάρα πολλέ περιπτώσει κατά τι οποίε δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα για να ενεργοποιηθεί μια έρευνα και έγινε ανάλυση κινδύνου και είπαμε ότι χρειάζεται. Είναι σημαντική αυτή η έρευνα και πολλέ φορέ επομένω εγκαταλείφθηκαν κάποιε επιχειρήσει γιατί έγινε μια τέτοια ανάλυση κινδύνου που οδηγούσε στην εγκατάλειψη. Και τελικά έγινε το κακό. Άρα, παρακάτω. Σε κάποια φάση είπαμε να δούμε κατά πόσον ε, καταλαβαίνουν οι δικαστέ τι γίνεται στις υπηρεσίες πληροφοριών. Να σας πω κάτι που μου συνέβη προσωπικά. Διορίστηκα στο νομικό τμήμα τη υπηρεσία πληροφοριών σε μια ταραγμένη εποχή. Υπήρχαν προβλήματα στις υπηρεσίες. Κάποιο είχε λιποτακτήσει απόστατη τέλο πάντων προς τους ε, που πάει στους, στους, Αλέξανδρου πήγε στους Ρώσους, κάποιος άλλος έγραψε μονεύματα και έλεγε σημεία και τέρατα. Τέλος πάντων ε, θα έπρεπε εμείς τώρα να δούμε τι θα κάνουμε ως νομικό τμήμα, ως νομική υπηρεσία. Και έλεγε ο νομικός σύμβουλος ότι δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις ούτε σε ένα χρόνο τι γίνεται στην υπηρεσία. Μου πήρε τρεις μέρες ακριβώς για να καταλάβω τι γίνεται στην υπηρεσία, πώς λειτουργεί το επίπεδο διαβάθμισης που υπήρχε για τις πληροφορίες. Οπότε, ένας έμπειρος δικαστής μπορεί να σταθμίσει τα αποδεικτικά στοιχεία, μπορεί να σταθμίσει αν έχουν κατα, καταπάτηση δικαιωμάτων, αλλά δε, αν θα καταλάβει την υπηρεσία, αυτό μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει, γιατί η δουλειά του είναι να υποβάλει ερωτήματα. Τώρα, τελευταίο, είχαμε διάφορες ε, παρατηρήσεις σε σχέση με το πώς η μία υπηρεσία παρακολουθεί την άλλη. Και σε σχέση με τις γερμανο-βρετανικές σχέσεις. Δεν ήρθα εδώ για να συζητήσω τα πολιτικά θέματα, γιατί αυτό είναι πολιτικό θέμα. Άμα κάποιες χώρες φοβούνται ότι τις κατασκοπεύουν, ε, ας πάνε να τα βρουν με τη χώρα που τις κατασκοπεύει. Ή ας πάνε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχει ακριβώς ε, Διασπάνε θεωρεί ότι παραβιάζονται τα ατομικά του δικαιώματα. Έχει γίνει αυτό ει βάρο του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, αυτή νομίζω είναι η επιτροπη ανθρωπινων δικαιωματων αν καποιο θεωρει οτι δεν τα ατομικα δικαιωματα εχει γινει αυτο εις βάρος του ηνωμενου βασιλειου αυτη νομιζω ειναι η λυση Και εδώ θα βάλω τελεία. Thank Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ όλους για όλες τις ε, ερωτήσεις που κάνετε. Ε, ε, έχω την εντύπωση ότι λίγο έχουμε καθυστερήσει, αλλά θα το καλύψει, θα καλύψει τη διαφορά ο αγαπητός φίλος Κλόντ Μωράης. Ευχαριστώ. όλους τους ομιλητές ε, για τις παρεμβάσεις τους και τις ερωτήσεις. Ε, έχουμε, ε, ζήτησαν πολύ να μιλήσουν παρότι ήδη είχαμε ακούσει τα μέλη του πάνελ. Αυτό δείχνει πόσο σας ενδιαφέρει το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε όπως προβλέπει το πρόγραμμά μας. Γι' αυτό το τμήμα της συζήτησης, επειδή είναι προφανές ότι θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα του ελέγχου των υπηρεσιών πληροφοριών, παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης. Ε, στην πράξη είστε και ειδικοί, ξέρετε πολύ καλά τα ζητήματα που τίθενται. Ε, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές του πρώτου τμήματος. Θα κάνουμε ε, μια μικρή διακοπή, ένα λεπτό, μέχρι να αλλάξουν τα μέλη του πάνελ. Ένα λεπτό διακόπη ε, μόνο για να αλλάξουν τα μέλη του πάνελ, παρακαλώ. Colleagues, if, um, if we want to get seated, we can, we can, uh... Παρακαλώ συνάδελφοι καθίστε για να μπορέσουμε να ξαναρχίσουμε. Στις 12.30 θα φάμε. The sooner we can... Uh, Όσο το δυνατόν συντομότερα ε, αρχίσουμε, τόσο γρηγορότερα θα φτάσουμε στο γεύμα. Please take your seats. Thank you. Okay. Let's get started. Thank you. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ιαν Κάμερεν από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, ο καθηγητής Κάμερον, καθίστε παρακαλώ και προσέξτε, θα σας πω, θα ακούσουμε την παρουσίαση της έκθεσης της Επιτροπής Βενετίας για το 2015 από πλευράς του καθηγητή Κάμερον. Θα του ζητήσω να μιλήσει 10 λεπτά, διότι βλέπω ότι έχετε ζεσταθεί τώρα και είστε έτοιμοι να κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις. Οπότε θα ήθελα να είναι διαδραστική η συζήτηση. Γίνεται σε 10 λεπτά, 12 ε. Αυτοί οι ακαδημαϊκοί πάντοτε θέλουν να, να υπερβαίνουν το χρόνο τους. Τέλος πάντων, πάνω κάτω 10 λεπτά σας παρακαλούμε. Και μετά θα ακούσουμε τον Δόκτρα Μάριο Οτχάιμερ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ τους διοργανωτές για τη σημερινή πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Διακόπτει ο κύριος Μωρές. Όσοι θέλουν να κάνουν πηγαδάκια, παρακαλώ να σταματήσουν. Δεν συνηθίζεται αυτό η διμερή συζήτηση μέσα στην αίθουσα. Ε, μπορείτε, μπορείτε να ε, μιλάτε ψιθυριστά, αλλά όχι όρθιοι. Δεν, δεν ε, ήθιστε στο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, εγώ θα σας παρουσιάσω την ε, επικαιροποίηση του 2015 για την έκθεση του Συμβουλίου της Βενετίας. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ξέρετε ότι είμαστε συμβουλευτικό σώμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και θεσμός του Διεθνούς Δικαίου το 2007 εξεπώνησε μια έκθεση η Επιτροπή της Βενετίας και εξακολουθεί να είναι σημείο αναφορά, αν θέλετε, σε αυτό το τομέα για τις βέλτιστες πρακτικές ως προς την λογοδοσία για του, τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών ε, ε, σε συνδυασμό με τον δικό εκπρόσωπο για την τρομοκρατία του ΟΗΕ και άλλους διεθνείς φορείς. Ε, πιστεύω ότι η Επιτροπή της Βενετίας ε, παραμένει το σημείο αναφοράς για τις βέλτιες πρακτικές. Λοιπόν, επικαιροποίηση το 2015. Ε, το σημείο εστίαζης είναι οι πληροφορίες σημάτων και εγώ ήμουν εισηγητής. Εξηγούμε τι είναι αυτό, τι είναι οι πληροφορίες σημάτων. Εξηγούμε γιατί μέχρι στιγμή δεν έχουν υπαχθεί σε επαρκείς εξωτερικούς ελέγχους και εξηγούμε επίσης πως το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χειρίζεται και προσαρμόζεται σε αυτές τις πληροφορίες σημάτων. Βλέπουμε τις ε, ε, βέλτιστες πρακτικές για στην ρύθμιση αυτών των πληροφοριών. Ε, συναντήσαμε πολύ σημαντικές δυσκολίες σε σχέση με την έκθεση του 2007, ε, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν ήδη ε, συστήματα σε διάφορα κράτη-μέλη, σε κάποια περίπτωση σε όλα, Ολλανδία, Βέλγιο, Σουηδία, εκεί οι εθνικές αρχές έχουν τέτοια συστήματα, στην Νορβηγία επίσης και όλα λειτουργούν εύρυθμα. Όμως ε, δύσκολα μπορούμε να βρούμε καλά μοντέλα για τις πληροφορίες σημάτων. Υπάρχουν δύο βασικά μοντέλα, το σουηδικό και το γερμανικό που δουλεύουν ιδιαίτερα καλά, αλλά και το αμερικανικό μετά την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας και αυτό παρουσιάζει ε, ενδιαφέρον. Το σημαντικό είναι να τονίσουμε το εξή. Όπως οι σημαντικές πρακτικές είναι ε, διαπαιδαγωγικού χαρακτήρα και ενθαρρύνουν τους άλλους να τις υιοθετούν, ε, ε, οι κακές αντίστοιχα πρακτικές μπορούν να ασκήσουν κακή επιρροή. Και το παρατηρούμε αυτό και στο πεδίο των υπηρεσιών πληροφοριών. Με το παράδειγμα των Γάλλων που απομακρύνονται από τους ε, δικαστικούς εισαγγελείς ε, και υιοθετούν το αμφιλεγόμενο και και ύποπτο θα έλεγα αγγλοσαξονικό μοντέλο. Ε, επίσης, ταυτόχρονα βλέπουμε μεγάλη επέκταση των κονδυλίων για τις πληροφορίες σημάτων μετά τις επιθέσεις 10 Σεπτεμβρίου. Όπως βλέπουμε, η βασική δικλίδα ασφαλείας για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα είναι ο επαγγελματισμός και η ακαιρεότητα των ίδιων των υπηρεσιών πληροφορίας. Και επειδή τώρα ε, πολλαπλασιάζονται οι πόροι, αν αυτό συνδυαστεί με πολιτική πίεση για να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα τότε, Ποιο είναι το αποτέλεσμα, απομακρύνεται από τους ελέγχους ε, η υπηρεσία πληροφοριών και βγαίνουν καουμπόιδες και ούτω καθεξής. Χρειαζόμαστε έλεγχο, το συμφωνήσαμε, δεν χρειάζεται να σου το εξηγήσω γιατί, διότι ε, δεν πρόκειται για παρα... παρακολούθηση της συμμόρφωσης ε, με τις εκείμενες διατάξεις, όμως αντικαθιστά τον έλεγχο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που απουσία του ελέγχου καλύπτει αυτό το κενό. Όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί στην περίπτωσή μας και θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί ε, χωλαίνει ε, αυτός ο τομέας της ε, ε σημάτων. Ε, όλα αυτά μπορείτε να δείτε σε λεπτομέρειες στην παρουσίασή μου που θα σας δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επίσης οι εκθέσεις 2007 και 2015 είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο μας. Υπάρχουν λοιπόν περιορισμοί ως προς ε, τις υπηρεσίες. Ε, πρώτα απ' όλα η εντολή. Δεύτερον, τα όρια που πρέπει να τηρηθούν προτού μπορέσει να αρχίσει συλλογή πληροφοριών, μια υπηρεσία πληροφοριών σημάτων και τρίτον οι απαιτήσει που υπάρχουν για τους μηχανισμούς αποκλεισμού μη, σημαντικών, μη σχετικών πληροφοριών και τέλος συμμόρφωση, παρακολούθηση συμμόρφωσης και έλεγχος της ε, ε, συμμόρφωσης για τα άνωθη στοιχεία. Θα πρέπει να αρχίσουμε λοιπόν με την εντολή. Η εντολή της υπηρεσίας είναι ουσιαστικά η εντολή ε, της υπηρεσίας ελέγχου. Δηλαδή, δίνεται ε, ε, την ε, υπηρεσία την εντολή να ε, συλλέγει πληροφορίες που έχουν σημασία για την τρομοκρατία ή για τις εξωτερικές υποθέσεις, ε, τότε θα θεωρηθεί ως κεκτημένο ότι έχουν πλέον τη δυνατότητα να συλλέγουν μαζικά στοιχεία σε σχέση με αυτούς τους τομείς, διότι πλέον έχουν την εντολή. Ε, στην πρωτογενή νομοθεσία πρέπει ε, να προβλεφθεί η σχετική διάταξη και ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να νομοποιηθεί για κάτι τέτοιο. Εάν υπάρξει μια διάταξη μέσα σε ένα καταστατικό, παρόλα αυτά εξακολουθεί να ισχύει η νομοθεσία και το προσωπικό είναι αυτό που εφαρμόζει την νομοθεσία νομοθεσία. Ε, Επίση, στι υπηρεσίε πληροφοριών οι νομοθετικέ διατάξει πρέπει να μετατραπούν σε λογισμικά. Ε, και, δηλαδή, κατοχυρώνουν διακαιρότητα μέσα από νομοθετικέ διατάξει και αυτέ οι νομοθετικέ διατάξει πρέπει να μετατραπούν σε ε, λογισμικά και στη συνέχεια αναλυτέ, υπάλληλοι, ε, θα εξάγουν τα στοιχεία μέσω του λογισμικού και θα τα αναλύσουν. Έτσι βλέπετε την αλυσίδα. Ε, ένα βασικό ζήτημα που μας απασχολήσει και αργότερα είναι ο τόπος διαμονής ε, και ε, η ηθαγένεια. Αν υπάρχει ηθαγένεια ή όχι και αν είναι ο τόπος διαμονής μόνιμος ή όχι για το άτομο που υπάγεται σε έλεγχο. Πρέπει να γίνει δεκτό ότι υπάρχει ιδιωτική σφαίρα και κατοχυρωμένα δικαιώματα ακόμη και για αλλοδαπούς ε, που δεν έχουν ε, μόνιμο τόπο διαμονής ε, στη χώρα. Όλες οι χώρες που είναι, είναι συμβαλόμενα μέρη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν δεχθεί αυτό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα έχουν προνομιακή μεταχείριση αυτές οι δύο κατηγορίες. Το αμερικανικό μοντέλο είναι σημαντικό γιατί μας δείχνει ότι δεν λειτουργεί ένας αμυγός κοινοβουλευτικός έλεγχος και έτσι συγκροτήθηκε ένα ανεξάρτητο ε, σώμα το οποίο ε, ασχολείται με την παρακολούθηση των υπηρεσιών πληροφοριών και την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας ακριβώς για να παρακούσει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ε, και μαζί με το δικαστήριο αυτός ο εθνικός φορέας προσφέρει ένα σχετικά καλό σύστημα ελέγχου στη ΣΥΠΑ. Όμως εστιάζουν περισσότερο στην προστασία των Αμερικανινών πολιτών και όχι ε, των υπολείπων στον υπόλοιπο κόσμο. Επιπροσθέτως ε, δεν έχει αρμοδιότητα το δικαστήριο ε, δικαιοδοσία στον τομέα των αμυγός αλλοδαπών πληροφοριών. Δεν μιλάμε για τις επικοινωνίες ανάμεσα στους Αμερικανούς και πολίτες σε τρίτων χωρών, αλλά ανάμεσα σε Γάλλους και Βρετανούς υπηκόους παραδείγματος χάρη γι' αυτό. Και ε, πρόκειται για μια διαφορετική εκτελεστική εντολή, ένα διάταγμα το 1233 που διέπει τις επικοινωνίες μεταξύ αλλοδαπών ε, και άρα ε, δεν εμπίπτει στην ε, δικαιοδοσία του δικαστηρίου ούτε και του εθνικού φορέα. Περάσω τώρα στην υπηρεσία πληροφοριών σημάτων. Να το πω απλά. Υπάρχουν δύο ε, λόγοι ε, δομικού χαρακτήρα που εξηγούν γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά ένα, λεπτά, ένα λεπτό να, να σας πω ότι υπάρχουν και σοβαρές τεχνικές ε, δυσκολίες, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να προσφύγουμε σε εξωτερική πραγματογνωμοσύνη. Δεν είναι το βασικότερο πρόβλημα. Δεύτερον, οι, οι βουλευτές πρέπει να βρουν και χρόνο να το κάνουν και το είπε ο κ. Σπυρακέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ο χρόνος, διότι πρόκειται για μια προϊούσα διαδικασία. Δεν μπορείτε να έρχεστε μία φορά στους πόσους μήνες και να το συζητάτε. Είναι μία διαρκής ε, πάγια διαδικασία και το ίδιο πρέπει να γίνεται και με τον έλεγχο ή τουλάχιστον να είναι τακτικός ο έλεγχος. Πέραν αυτού υπάρχει και το θέμα του δίκτυου. Πρόκειται για ένα δίκτυο και το ανέφεραν οι Γερμανοί συνάδελφοι ότι υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία ε, στο ζήτημα, δηλαδή το να δοθούν ε, διαβαθμισμένες πληροφορίες σε ένα κοινοβουλευτικό σώμα είναι κάτι πολύ δύσκολο διότι αποκαλύπτονται άλλες δραστηριότητες του δικτύου των ε, αυτών των υπηρεσιών δηλαδή με τις οποίες συνεργάζεται η ελεγχόμενη υπηρεσία πληροφοριών και άρα χρειάζεται ειδική εξέταση των πληροφοριών που θα κοινοποιηθούν. Πέραν αυτού, και το είπαμε, η, πληροφορία σημάτων ε, μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εποπτεία παραδοσιακά ήταν δουλειά του δικαστικού σώματος στην παραδοσια... στον παραδοσιακό διαχωρισμό εξουσιών. Αυτό σημαίνει ότι είναι προβληματικό να δοθεί στο Κοινοβούλιο μια σχεδόν δικαστική εξουσία. Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα ε, ακριβώς λόγω της επιρροής που έχει πληροφορία σημάτων για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρώτον, η επιλογή των φίλτρων επιλογής και δεύτερον η απόφαση ε, των υπηρεσιών να διατηρήσουν, να διαγράψουν τις ε, πληροφορίες. Η πρώτη, το πρώτο είδος αποφάσεων λοιπόν σε σχέση με τα φίλτρα επιλογής δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι πολιτικού χαρακτήρα, είναι σχεδόν δικαστικού. Είναι μια απόφαση που προϋποθέτει εξισορρόπηση διαφόρων παραγόντων και χρειάζεται αρμόδιες φορές για να γίνει αυτό. Χρειάζονται δικαστές που θα εργάζονται σε αυτό το φορέα και μπορεί να έρθουν και άλλοι που είναι ειδική σε μεθόδους ε, συλλογής ε, ή πληροφοριών ε, ή ειδικοί για εξωτερικά ζητήματα κτλ. Γι' αυτό και έχουμε υβριδικού τύπου σώματα στην Γερμανία και στη Σουηδία. Υπάρχει μεικτή σύνθεση λοιπόν σε αυτό στους φορείς, ε, αλλά παρόλα αυτά ίσως δεν είναι δυνατόν αυτό γιατί υπάρχει όπως είπαμε παραδοσιακό διαχωρισμός των εξουσιών. Πάντως ε, και η Γερμανία και η Σουηδία έχουν υιοθετήσει αυτό το μοντέλο. Το δεύτερο είδος αποφάσεων, ε, δηλαδή διατήρησης ή διαγραφής δεδομένων, αυτό είναι ζήτημα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων και λαμβάνεται η απόφαση από το προσωπικό του φορέα που συνυπολογίζει διάφορους παράγοντε. Ε, και ιδιαίτερα προβληματικό είναι να αποφασίσουμε ποιε πληροφορίε ε, χρειάζεται η υπηρεσία. Πολλέ συλλέγονται γιατί μπορεί και να προκύψει ανάγκη, μπορεί και να χρειαστούν στο μέλλον αυτές οι πληροφορίες. Οπότε ε, πρέπει να ζυγίσουμε το συμφέρον του να διατηρηθούν οι πληροφορίες στην ίδια πλάστηγα με την ανάγκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ούτε αυτή είναι η απόφαση που πρέπει να λάβει μία ένα κοινοβούλιο, ένα κοινοβουλευτικό σώμα ε, είναι απόφαση ενός φορέα προστασίας των ανθρωπίνων δημονών. Πρέπει να εξετάσει τη βάση δεδομένων, να αναρωτηθεί για ποιο λόγο διατηρήσατε εσείς αυτά τα δεδομένα για το συγκεκριμένο άτομο. Δείξτε μου το ίχνος ε, που και την έγκριση, την αρχική. Δείξτε μου την απόφαση ε, στην οποία βασιστήκατε για να κάνετε μια εξισορρόπηση των διαφόρων παραγόντων. Χρειάζεται ανεξάρτητος σχεδόν δικαστικού χαρακτήρα φορέας που θα εποπτεύει ε, την ε, τις πληροφορίες σημάτων. Ε, έχω επίγνωση του ότι υπερβαίνω το χρόνο μου, όμως είναι σημαντικό να σας πω ε, το εξή. Θα, μου, θα στραφείτε τώρα και θα μου πείτε, μα ε, τι μπορεί να κάνει το κοινοβούλιο, δεν, ε, τι, τι απομένει για το κοινοβούλιο και φυσικά είναι σημαντικό το κοινοβούλιο να παρέμβει. Μόνο εκείνο μπορεί να αποφασίσει τους γενικούς κανόνες σε σχέση με το πώς πρέπει να συλλέγονται οι πληροφορίες, πώς θα ανταλλάσσονται με άλλους φορείς και οργανισμούς και μόνο το κοινοβούλιο θα έπρεπε να είναι σε θέση να αποφασίσει σε γενικό επίπεδο ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, ω στην την ασφάλεια. Δηλαδή ο στόχος συλλογή των ε, πληροφοριών μόνο το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει για τη χρηματοδότηση και για την ε, αποτελεσματικότητα άρα του συστήματος πληροφορία σημάτων και τέλος, και εδώ αναφέρθηκα συγκεκριμένα στο γερμανικό και σουηδικό μοντέλο, μπορεί να έχει ρόλο το Κοινοβουλίο σε σχέση με αυτό τον ανεξάρτητο ε, φορέα που συγκροτείται, μπορεί να διορίζεται και να λογοδοτεί το σώμα αυτό, ο φορέας αυτό στο Κοινοβούλιο ή μπορεί να συνδεθεί ε, με ε, διαφορετικούς τρόπους με το Κοινοβούλιο, όπως το γερμανικό G10. Το Κοινοβούλιο μπορεί να προσφέρει κίνητρα στο σώμα για να επιτελεί σωστά τα καθήκοντά του. Μπορεί επίσης να υπερασπιστεί τον φορέα αυτό εάν δεχθεί αδικαιολόγητη κριτική. Ε, μπορείτε λοιπόν <clears throat> να έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, μου δίνετε κι άλλα λίγα λεπτά για να μιλήσω για το δικαστικό σύστημα, δύο λεπτά. Δικαστική έγκριση. για τα φίλτρα επιλογή. Δεν είναι πανάκι αυτό, μιλάμε για τους δικαστές, όμως θυμηθείτε ότι έχουμε διαφορετικές δικαστικές παραδόσεις εδώ στην Ευρώπη και έχουμε διαφορετικά επίπεδα δικαστικής εξουσίας ε, ανά κράτος μέλος. Είναι σημαντικό λοιπόν ε, να συνειδητοποιήσουμε ότι Έχουμε όλοι τις παροπίδες μας και λειτουργούμε βάσει των εφισταμένων συστημάτων. Τι είναι σημαντικό τώρα, ότι χρειαζόμαστε και τα δύο. Δεν αρκεί η δικαστική έγκριση, ούτε και αρκεί ε, να έχετε ενσωματωμένους στο φορέα δικαστές. Ε, ο κύριος Μπέκ μας μίλησε για τον γαλλικό σύστημα. Λοιπόν, το πρόβλημα αυτού του συστήματος είναι ότι ε, δεν είναι αποσπασμένοι πλέον οι δικαστές ενσωματώνται στο σύστημα το οποίο υποτίθεται ελέγχουν. Ε, δεν είναι πλέον ανεξάρτητη. Γι' αυτό σας είπα ότι χρειάζεστε μια σχεδόν ε, ή μη δικαστική έγκριση για να λειτουργήσει ο φορέας και για να συνδεθεί αυτό με, την, ε, με το follow-up τη συνέχεια που δίνεται. Δεν ξέρει πάντοτε ε, η δικαστική εξουσία πώς χρησιμοποιούνται οι εντολές και οι εγκρίσεις που δίνει, άρα πρέπει να υπάρξει μια σχέση, να συνδεθεί δηλαδή η έγκριση με το follow-up και στο follow-up θα πρέπει να υπάρχει έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα δεδομένα. Ε, δεν μπορεί να ε, ε, ισχύσει ο κανόνας για τα δεδομένα του τρίτου μέρους, δηλαδή χρειάζονται θεματικές μελέτες και μελέτες για την εξαγωγή δεδομένων όπως γίνεται στο σουηδικό και γερμανικό μοντέλο. Υπάρχει άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Δεν χρειάζεται να πάρουν τηλέφωνο και να πούνε έρχομαστε σε δύο εβδομάδες και άρα δίνουν το χρόνο στο, στον αρμόδιο φορέα να προετοιμαστεί και να μαζέψει τα πτώματα ε, και να καθαρίσει το χώρο. Όχι, έχουν άμεση πρόσβαση ε, στη βάση δεδομένων. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί ε, τρόποι, πολλές αναλλακτικές λύσεις. Θα ήθελα να κλείσω όμως την παρουσίασή μου λέγοντας πως είναι δύσκολο σε τόσο περιορισμένο χρόνο να αναφερθώ ε, σε όλα τα σημεία αυτού του περίπλοκου ζητήματος. Το πιο σημαντικό από πλευρά Επιτροπής Βενετίας ε, είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρέπει να εξαφανιστεί η πληροφορία σημάτων επειδή δεν μας αρέσει, ούτε πρόκειται οι υπηρεσίες πληροφοριών ε, να αποδιαρθρώσουν τις υπηρεσίες πληροφορίες σημάτων, αλλά ή μπορούμε να έχουμε μια χαλαρή ρύθμιση και έλεγχο ή το αντίθετο να υπάρχει ε, στενός έλεγχος ε, και πολύ συγκεκριμένη ρυθμίση και αυτό θα έπρεπε όλοι να επιδιώκουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ καθηγητέ Κάμερον. Θα ανεβάσουμε με την άδειά σας στο διαδίκτυο την παρουσίασή σας. Δεν ήθελα να σας διακόψω γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, ιδιαίτερα αυτά τα τελευταία ε, αμφιλεγόμενα ζητήματα που ε, αναφέρατε. Θέλω όμως να ε, γίνει και συζήτηση γι' αυτό κύριε όταν εσείς ε, από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εσείς μπορείτε να ε, τηρήσετε αυτή την, την το, το, όριο των 10 λεπτών που σας έστειλα. Θα μας παρουσιάσετε τη συγκριτική μελέτη του FRA σχετικά με το δημοκρατικό έλεγχο είστε επικεφαλή του Τμήματος Κοινωνία των Πληροφοριών του οργανισμού που εκπροσωπείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας ε, παρουσιάσω τα προκαταρκτικά ε, πορίσματα της μελέτης που διεξήχθη έπειτα από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σχετικά με τα ένδικα μέσα και τις ε, εγγύησει για την ε, διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Going for sake of time. Uh, anyway, you've received here a uh, background note on the Λοιπόν, λάβατε ένα σημείωμα στο οποίο μπορείτε να ανατρέξετε αν θέλετε και περισσότερες πληροφορίες. Το χρόνο που μου δόθηκε θα επικεντρωθώ σε τρία βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την επιτήρηση και συγκεκριμένα την προστασία της ιδιωτικότητας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρώτα απ' όλα, να σας μιλήσω για τα πρότυπα. Το, το ζήτημα των ένδικων μέσων που σχετίζονται αυτά τα δύο θέματα βεβαίως με την επιτήρηση και την εποπτεία και βεβαίως με χαρά θα δεχτώ και τα ερωτήματά σας μετά την παρουσίασή ε, Εδώ βλέπετε τα τρία βασικά ζητήματα που θα ήθελα να συζητήσουμε, να σας παρουσιάσω δηλαδή. Πρώτον, το πεδίο της ε, επιτήρησης ε, παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από μυστικότητα ενώ ε, και παρά το γεγονός ότι το έργο των μυστικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι μυστικό προφανώς θα πρέπει ωστόσο να διέπεται από σαφές νομικό πλαίσιο. Επίσης, τα άτομα, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένομη προστασία. Και τρίτον, τα συστήματα εποπτείας διαφέρουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως ε, η ανεξαρτησία των φορέων, είτε πρόκειται για δικαστές είτε για εμπειρογνώμονες, ε, σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι ε, θα χαρακτηρίζεται και από το στοιχείο της λογοδοσίας. Να ξεκινήσω με τα πρότυπα. Ακούσαμε πολλά και στην παρουσίαση του κυρίου Μπρίκφορντ. Εδώ βλέπετε σε απλουστευμένη μορφή τα πρότυπα που προβλέπονται με βάση της, ε, ε, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Χάρτα. Ο κύριος Μπίκφορντ επικεντρώθηκε στην ομολογία και την ε, νομοθεσία που σχετίζεται με την επιτήρηση. Το δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι η επιτήρηση δεν μπορεί να, είναι, να βασίζεται σε, ε, στην τυχαιότητα. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ε, διατύπωση προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Επίσης, υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχουν και εγγύησει με δύο στοιχεία. Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί εποπτείας και επιτήρησης και δεύτερον, θα πρέπει να προσφέρονται ε, κατάλληλα ένδικα μέσα στους πολίτες. Ο ειδικό ε, εισηγητής Μπεν Έμεσον του ΟΗΕ πρόσθεσε σε αυτά τα δύο και δύο ακόμη σημεία. Πρώτον, ότι η επιτήρηση θα πρέπει να σέβεται τις αρχές της αναγκαιότητας και της ε, αναλογικότητας. Δηλαδή θα πρέπει να, αιτιολογ, να, είναι να αιτιολογούν τα κράτη τα μέτρα που λαμβάνουν, αλλά και να αποδεικνύουν ότι τα μέτρα αυτά είναι αποτελεσματικά. Δεύτερον, το είπε και ο Ίεν Κάμερον πριν από λίγο, ε, η ιδιωτικότητα ως αρχή αφορά όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους ή την εθνικότητά τους. Εδώ μιλούμε για ελάχιστα πρότυπα. Ε, ελάχιστα πρότυπα που καταρτίζονται σε, εθνικό, σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς μπορούν ε, αυτά τα πρότυπα να ε, εφαρμοστούν υπό το φως των αποκαλύψεων του Edward Snowden και δουλειά της Επιτροπής Βενετίας είναι να αποφανθεί και επ' αυτού του ζητήματος ενώ περιμένουμε και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και δεύτερον, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς τα πρότυπα αυτά μπορούν να αναπτυχθούν και να προσαρμοστούν στα εθνικά δεδομένα. Εδώ σας ε, ε, παρουσιάζω τα ένδικα μέσα που ε, ισχύουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αλήθεια ότι οι πολίτες μπορούν να προσφύγουν στους, ε, στα δικαστήρια. Ωστόσο, αποδεικνύεται από την εμπειρία μας ότι οι πολίτες δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτές τις μακροχρόνιες διαδικασίες που είναι αναγκασμένοι να ακολουθούν όταν κανείς προσφεύγει στα δικαστήρια. Επίσης, δηλαδή θα πρέπει να ε, υπάρχουν και δικαστές οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα εμπιστευτικά έγγραφα και γι' αυτόν τον λόγο πολλά κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει τη σύσταση ειδικών ε, δικαστηρίων για ζητήματα σχετικά. Άρα πολλοί πολίτες έχουν την εναλλακτική λύση να προσφύγουν σε μη δικαστικού χαρακτήρα φορείς. Και εδώ βλέπετε εδώ τις διάφορες επιλογές που έχει κανείς, κοινοβουλευτικές επιτροπές, ε, εκτελεστικούς φορείς κτλ. κτλ. Το πρόβλημα με, τα, με τους μη δικαστικούς φορείς είναι ότι πολλές φορές έχουν πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες μόνο τα μισά κράτη-μέλη έχουν ε, φορείς που μπορούν να λαμβάνουν και αποφάσεις. Εγώ θα επικεντρωθώ τώρα στο ζήτημα της εποπτείας, όπως είναι και το θέμα της, διάστη, της διάσκεψής μας. Εποπτεία είναι η λογοδοσία για τη λήψη αποφάσεων. Και εδώ προσπαθώ να σας δείξω ποιοι είναι οι παράγοντες που διαδραματίζουν ρόλο στο ε, σύστημα. Εδώ μπορείτε να δείτε τους ε, μηχανισμούς λογοδοσίας και παρότι υπάρχουν πολλές φορές δεν προβλέπονται από την ε, νομοθεσία τα μέτρα που, μπορεί που μπορούν να λάβουν. Φυσικά οι μη κυβερνητικές οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο και οι αποκαλύψεις Snowden το 2013 απέδειξαν πόσο σημαντικές είναι οι μη κυβερνητικές, οργανω... Ε, οργανώσεις. Επίσης, σε πολλά κράτη-μέλη οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις υποβάλλουν ε, αγωγές που σε πολλές περιπτώσεις ακόμη εκκρεμούν. Λειτουργούν δηλαδή ως ε, ως ένας ε, μηχανισμός διασφάλισης της νομιμότητας και όπως ε, αποδεικνύεται και σε σχετικές περιπτώσεις στη Γαλλία είναι πάρα πολύ σημαντικές οι μη, ε, κυβερνητικέ οργανώσεις όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας. Επίσης υπάρχει το, η Ευρωπαϊκή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την οποία πρέπει να τηρούν τα κράτη-μέλη. Τα επόμενα λεπτά θα επικεντρωθώ σε τρεις πιο δομημένους ε, φορείς επιτήρησης στα κράτη-μέλη. Ε, είναι η κοινοβουλευτική επιτήρηση αφενός ε, που ε, το αναφέραμε ήδη είναι επιφορτισμένη με την κατάρτιση των προτύπων την έγκριση των προϋπολογισμών ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσει για τις πληροφορίες σημάτων αλλά επίσης οι κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν και αρμοδιότητες διερεύνησης υποθέσεων υπάρχουν Δεύτερον, οι φορείς εμπειρογνωμόνων και οι δικαστικοί φορείς, εξάντε ή εξπόστ. Να περάσω τώρα στην έγκριση των ε, στοχευμένων μέτρων επιτήρησης, όπως ε, ισχύουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όπως αποδείχθηκε και από την συζήτηση πριν, είναι πολύ σημαντικό να ε, η επιτήρηση να διεξάγεται με νόμιμο τρόπο και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προβλέπεται συγκεκριμένο σύστημα. Σε περισσότερα από τα μισά κράτη-μέλη, ε, εισαγγελείς ή δικαστές εγκρίνουν τα μέτρα επιτήρησης. Στα άλλα μισά κράτη-μέλη αυτό, αυτός ο ρόλος αναλαμβάνεται από εμπειρογνώμονες ή από την κυβέρνηση. Και αυτό αφορά, ε, είναι μια, ε, αυτό προβλέπεται και στην Ευρωπαϊκή Χάρτα. Υπάρχουν και δύο κράτη-μέλη στα οποία δεν απαιτείται καμία έγκριση. Και να σας επισημάνω μια υπόθεση που εκρεμεί ε, στο δικαστήριο εδώ, Ζάμπο, εναντίον Ουγγαρία, που εκκρεμεί ακόμη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όσον αφορά την έγκριση των πληροφοριών σημάτων, νομίζω το είπε και ο, ο κύριος Κάμερον, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ σε αυτή τη διαφάνεια μπορείτε να δείτε τις διάφορες πρακτικές που ακολουθούνται σε τέσσερα κράτη-μέλη όπου υπάρχει λεπτομερής νομοθεσία που διέπει τις πληροφορίες σημάτων. Όσον αφορά τον, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος ε, διεξαγωγής του ελέγχου. 24 κράτη-μέλη, σε 24 κράτη-μέλη τα κοινοβούλια ε, επιτηρούν τις μυστικές υπηρεσίες, έχουν δηλαδή κάποιες αρμοδιότητες. Ωστόσο, ε, ε υπάρχουν ε, κάποιες βασικές αρμοδιότητες, υπάρχουν και κάποιες ενισχυμένες αρμοδιότητες όσον αφορά την υποδοχή καταγγελιών και να περάσουμε στα ειδικά, στους ειδικούς, ε, ειδικούς φορείς εμπειρογνωμόνων. Τέτοιου είδους ε, φορείς έχουν συσταθεί σε 14 κράτη-μέλη και μάλιστα κάποια κράτη-μέλη έχουν συστήσει και περισσότερο από ένα τέτοιο φορέα. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των φορέων, των σωμάτων, είναι θα πρέπει να έχουν ε, τις απαραίτητες το είπε και ο κύριο Κάμερον όσον αφορά την εντολή του. Αλλά επίσης θα πρέπει να έχουν και τους κατάλληλους πόρους αλλά και να λειτουργούν ανεξάρτητα. Και μία και μιλούμε για την ε, προστασία της ε, μας ενδιαφέρει να δούμε πώς ε, οι αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στον ε, τομέα και στο πεδίο της ε, επιτήρησης. Εδώ σε αυτό το χάρτη μπορείτε να δείτε με ποιον τρόπο τα 28 κράτη-μέλη και οι 28 αντίστοιχες αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορούν να συνεργαστούν με άλλους μηχανισμούς επιτήρησης. Βλέπετε εδώ από το χάρτη ότι υπάρχει μια σειρά από λύσεις στις οποίες μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες από μια πλήρως ε, εξοδοτημένη αρχή έως και αρχές με περιορισμένες εξουσίες, δηλαδή που αντιμετωπίζουν ε, εμπόδια σε σχέση με τις ε, επαφές τους με τις μυστικές υπηρεσίες και υπάρχουν και μια τρίτη κατηγορία εκείνων των ε, χωρών που δεν έχουν καθόλου ε, ε, αρμοδιότητες και εξουσίες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ το διάγραμμα που βλέπετε τώρα, το οποίο δεν θέλουμε απλά να αποτυπώνει την ποικιλομορφία που υπάρχει στα κράτη-μέλη, αναδεικνύονται και κάποια ερωτήματα μέσα από αυτό το διάγραμμα. Τι συμβαίνει στα τέσσερα κράτη-μέλη που έχουν σώμα εμπειρογνωμόνων και αρχή προστασία ε, προσωπικών δεδομένων ή αντίθετα τι συμβαίνει στα πέντε κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, ε σώμα εμπειρογνωμόνων ούτε αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων με πλήρε εξουσίες. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν θα απαντήσει η δική μας συγκριτική μελέτη γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο, περισσότερη έρευνα και έργο ε, επιτόπου. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Να προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε δηλαδή ε, να διεξάγουμε έρευνα επιτόπια. Στο δεύτερο εξάμεινο φέτος θα ε, προσπαθήσουμε να κάνουμε συνεντεύξεις με ε, εμπειρογνώμονες, με κοινοβουλευτικές επιτροπές, τους βασικούς φορείς δηλαδή σε εθνικό επίπεδο. Με εκείνου δηλαδή τους φορείς με τους οποίους θα θέλαμε να συζητήσουμε και τα πορίσματά μας. Δεν ε, υποτιμώ τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε σε καμία περίπτωση, αλλά νομίζω παρόλα αυτά ότι είναι ο μόνος τρόπος και ο μόνος δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να απαντήσουμε και στα αιτήματα που μας έχει υποβάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα τα βασικά ζητήματα θα ήθελα να, ε, επαναλάβω. Το νομικό πλαίσιο είναι μια προϋπόθεση και μόνο και θα πρέπει πάντοτε να επικαιροποιείται με βάση τις εξελίξεις. Ή θα πρέπει με, κάποιον, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να ε, υπάρχουν ε, ένδικα μέσα στα οποία μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες και θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα ε, επιτήρησης αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος στον εκπρόσωπο. Μπορούμε να αφήσουμε αμέσως στις ερωταπαντήσεις. Έχουμε ήδη τον κατάλογο των αγορητών. Οπότε συνάδελφοι, συμπλώστε αυτό το έντυπο και πέστε μας αν θέλετε, αν ήδη δεν το έχετε πράξει. Παρακαλώ να έχουν προτεραιότητα τώρα οι συνάδελφοι που δεν υπέβαλαν ερωτήσεις μέχρι τώρα. Ε, Ρουίς, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Ρουίς, υποβάλλατε την ερώτησή σας. Sorry. I'm, I, I'm not to this straight with you? Mr. Ruiz, are you hearing this at all? Κυρία Ρουίς, επιμένει ο Πρόεδρος. Θέλετε να υποβάλλετε ερώτηση. Yeah. Please go ahead. Por supuesto, perdón. Βεβαίω, βεβαίω και συμπαθάτε με πρόεδρε. <laughs> Συγγνώμη, δεν κατάλαβα ότι απευθύνεστε σε μένα. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ό,τι είπαν οι συγκητέ και οι προηγούμενοι και αυτοί. Όταν μιλούμε για υπηρεσίες ε, ασφάλειας, τότε μιλούμε για διαφορετικά πράγματα ανάλογα με τη χώρα. Οι δε τεχνολογικές εξελίξεις σε έναν κόσμο που συνέχεια αλλάζει όπως ελέγχθη αφορούν το πόσο κανείς μπορεί να παρέμβει, να χειραγωγήσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα. Άρα Τώρα τα πράγματα είναι πιο έντονα παρά ποτέ και στη δική μας χώρα ανήκαθεν έπρεπε να πασχίσουμε για να ανασχέσουμε επί δεκαετίες την τρομοκρατία. Οπότε και τα θέματα πληροφορίας αλλά και τα θέματα τα αστυνομικά τα χειριστήκαμε ακριβώς ως χώρα για να δούμε πώς θα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Αλλά επίσης για να μπορέσουμε να περιχαρακώσουμε και τα όρια των δραστηριοτήτων αυτών. Έχουμε ένα ειδικό δικαστήριο. Αυτό λέγεται εθνικό δικαστήριο. Οι δικαστές που εκεί υπηρετούν είναι εξειδικευμένοι σε θέματα οργανωμένου εγκλήματο αλλά και τρομοκρατίας. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Δεν θα πρέπει απομονωμένα να αντιμετωπίζουμε τις υπηρεσίες ασφαλείας. Θα πρέπει να τι αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την συνήθι δράση της αστυνομίας. Γιατί υπάρχει τη τρομοκρατία και ο εγκλήματο. Να, να τα πασάρουμε στις υπηρεσίες πληροφοριών και όχι στην αστυνομία εύκολη λύση. Οπότε πέραν των όσων ελέγχθησαν εδώ τώρα για την πρικοδότηση των υπηρεσιών όσον αφορά τις έρευνες, όσον αφορά τους εποπτικού ε, ελέγχους, θα πρέπει να δούμε ότι στο οργανόγραμμα ε, των αντιβιωτικών αρχών είναι συμπληρωματική δράση των μεν υπηρεσιών με τις δε, την, ε, την αστυνομία. Οπότε με τα μέσα που είναι διάθεσή μας είναι αναγκαιότητα στο να μπορούμε να δούμε το πώς θα υπάρχει κάποια κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι το οποίο στην αρχή της διαδρομής μας δεν το είχαμε. Επομένως, τι μπορεί να κάνει στην καθημερινή της δράση η αστυνομία, πώς μπορεί να αξιοποιήσει πρωτόκολλα και μέσα, τι ε, επιφυλάσσεται τελικά στις ε, υπηρεσίες πληροφοριών. Γιατί υπάρχουν κάποιοι συστημικά δίκτυα, συστημικά και όχι συγκυριακά. Οπότε έχουμε οργανωμένο έγκλημα και δρομοκρατία που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε όλο το τοπίο μαζί. Χρειαζόμαστε όλες τις πληροφορίες, όλα αυτά τα οποία εσείς μας είπατε που κάνουν οι υπηρεσίες αυτές. Άρα να δούμε σε σχέση με την αστυνομία. Πώς θα μπορέσουμε να υπάρχει συμβατή συνεργασία, συμβατή συνύπαρξη αυτών των υπηρεσιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν έφτακτα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Άρα Ας ε, καθορίσουμε και ας ορίσουμε τι θα πρέπει να κάνουν οι υπηρεσίες πληροφοριών και τι αστυνομία. Γιατί είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν είχαν τόση εξουσία υπηρεσίες πληροφοριών. Ποτέ δεν ε, ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα σε σχέση με τη δημοκρατία. Να, η πρόκληση του 21ου αιώνα. Επομένω, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι οι κατευθύνσει πώ θα το θα δώσουμε. Όλα αυτά θα πρέπει να διέπονται από η ισορροπία. Πρόεδρο. Ευχαριστούμε. Δεν ήταν ερώτηση αυτό που είπατε, πιο πολύ ήταν δήλωση, αλλά οι συνάδελφοι αν θέλουν θα τοποθετηθούν πάνω σε αυτό. Φραντς Πέρχαπ, από την Bundesrat, πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων. Κύριε Μπέρχαπ. Thank you. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, είχαμε μια εξεταστική επιτροπή στην Bundestag. Και προκύψει ότι η Αυστρία εμπλέκεται. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικός ισχυρισμός κατά μας για θέματα εσωτερικής εθνικής ασφάλειας και προστασίας. Άρα αυτό το ελάβαμε πολύ σοβαρά υπόψη. Και θέλω να ρωτήσω τους δύο συγκητές τι θα πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει από νομικής πλευράς στο μέλλον, τόσο ώστε να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα. Και να μην έχουμε διαρροή τέτοιων πληροφοριών προς τρίτους, όπως την υπηρεσία ασφαλείας τον είπα. Να δούμε πώς θα έχει πληροφορίες που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα-πρώτα. Και είναι δυνατόν να έχουμε παροχή πληροφοριών προς τις φίλες και φιλικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν σύντομος, λέει ο Πρόεδρος. Παρακάτω. Εύα Ζολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή. Μέχρι τώρα έχω δεν υπάρχει αυθεντική εποπτεία επί των υπηρεσιών. Και δεν έχουμε ακόμα συλλάβει το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. στη Γαλλία, μέχρι το 2007 είχαμε περίπου 6.000 ελέγχους διοικητικούς ετησίως. Και υπήρχε μια επιτροπή αρμόδια να εποπτεύει σε αυτές τις παρακολουθήσεις. Τώρα έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ακροάσεων και παρακολουθήσεων. Και ε, έχουμε τώρα κάποια επιτροπή από δικαστικούς η οποία ε, λειτουργεί διαλυπώντος. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Κάμερον από το Πανεπιστήμιο της Ουσάλα. Εσείς έχετε αναλάβει κάποιες μελέτες όσον αφορά την ασυμμετρία των μέσων. Από τη μια μεριά έχουμε τις υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ψηφίσει αποτελεσματικά μέτρα που τα κάνουν, τα ξέρουμε, αλλά είδαμε και με την ΕΝΕΣΑ την υπηρεσία των ΙΠΑ. Και έχουμε δεκάδες χιλιάδες στις ε, ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών και είπαμε ότι ε, έχουμε την υποπτία ε, από κάποιους λίγους που δεν γίνεται καν συνέχεια. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει γιατί τώρα έχουμε βρεθεί με το παλιό μοντέλο, το οποίο δεν επαρκεί, ήταν αλλιώ τότε τα πράγματα. Άρα θα πρέπει να μελετηθεί αυτή η ασυμμετρία. Έχετε κάποια πρόταση πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, Ευαλία Πρόεδρος. Και τώρα. Πώς έγινε ο Σάντζεθ από την Ισπανική Βουλή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία σκέψη για τους συναδέλφους από τα κοινοβούλια. Πριν μας μίλησε ο κύριος ε, Μπράκε για το τι γίνεται, ποιος είναι ο ρόλος των ε, βουλευτών και τα δικαιώματα των πολιτών και για το πόσο από την άλλη μεριά θα πρέπει να, να είναι υπηρεσίε αποτελεσματικέ. Να, που δούμε την ισορροπία. Όμω, ακριβώ όσο συζητήσαμε από την αρχή τη συνάντηση, αυτή που είναι υπέρ της ελευθερίας των υπηρεσιών θα πρέπει να είναι πολύ χαρούμενοι γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας αυτοπρισμός και αυτοπιθαρχία στους βουλευτές. Είναι σαν να αναγνωρίζουν το ότι δεν μπορούν ή δεν πρέπει να ε, ασκούν έλεγχο κοινοβουλευτικό επί των υπηρεσιών. Και επινοούνται όλες οι δικαιολογίες. ας πούμε να πριν από 25 χρόνια ότι θα πρέπει να ξέρει πώς δουλεύει το τηλέφωνο για να κάνει κάποιο είδους ε, παρακολούθηση είπε ε, και ο Ιταλός ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε κάποιον έλεγχο της προκοδότησης. και είπε, ο Τσέχος συνάδελφος είπε ότι ο έλεγχος των υπηρεσιών ε, γινόταν από πρώην πράκτορες, πρώην στελέχη. όλα αυτά είναι επιλήψιμα γιατί όπως έλεγε ο ίδιος τελικά το, το, το, το, ενδιαφέρον, αυτό που έχει για τους πολιτικούς είναι να μην σπηλωθεί το, το κόμμα τους. Εγώ όμως ως βουλευτής θεωρώ ότι αυτό που με καίει είναι τι γίνεται με τα δικαιώματα των πολιτών, γιατί το θέμα δεν είναι αν ε, υφίσταται κατασκοπή ή παρακολούθηση ένα κόμμα, το θέμα είναι να μην κατασκοπεύεται κανείς πολίτης. Επομένως, πρέπει να διαδραματίσουμε έναν ρόλο πολιτικό. Οι δικαστές να ελέγξουν να αδειοδοτούν, να ελέγχουν πολιτικά. Γιατί πρόκειται για ακόμα μία λειτουργία κυβερνητική. Να γίνεται ό,τι γίνεται με τις άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα είναι άλοθη και είναι επιχειρήματα έολα. Α, μας είπε και ο κύριος από την Επιτροπή της Βενετίας ότι είναι κάτι το πάρα πολύ σοφιστικέ, πάρα πολύ τεχνοκρατική κατάσταση, το επίπεδο δηλαδή των μέσων που έχουν, μα τι. Μα γιατί δεν καθόμαστε και να κουβεντιάζουμε στα κοινοβούλια για τα πυρηνικά κέντρα, χωρί να είμαστε πυρηνικοί επιστήμονε. Μα δεν είναι δυνατόν να έχουμε ω πρόφαση ε, την τεχνολογία για να μπαίνει τροχοπέδι στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν χρειάζεται τεχνική γνώση για να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ναι, μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητου δικαστέ και ανεξάρτητου εμπειρογνώμονε, αλλά δεν είναι δυνατόν εμεί να ερχόμαστε εδώ και να λέω ένα στον άλλο ότι εμεί απεμπολούμε το καθήκον μας του πολιτικού ελέγχου όσον αφορά τη δραστηριότητα των υπηρεσιών. Και αναφέρθηκε πολλές φορές σήμερα το πού μπορεί να υπάρχει έλεγχος. Όχι όπως έλεγε η Γαλλίδα συνάδελφος, περιπτωσιολογικά. Να γίνεται έλεγχος έστω και εκ των υστέρων όπως γίνεται παντού σε όλες τις υπηρεσίες. Όπως γίνεται με τον έλεγχο της αστυνομίας. Και εκεί υπάρχουν θέματα πολιτικά λεπτά. να μην βγει το συμπέρασμα από εδώ μέσα ότι δεν είμαι θα θέση να ασκήσουμε έλεγχο επί αυτών των υπηρεσιών όπως ελέγχουμε όλες τις υπόλοιπες και δεν μπορούμε και το αφήνουμε στους ε, κάποιους εμπειρογνώμονες και παίοντες. Μα τότε και οι πολίτες θα πρέπει οι ίδιοι να κάτσουν και να προστατεύσουν τον ιδιωτικό τους τα δικαιώματά τους να δεν το κάνουν οι βουλευτές. Thank Σας ευχαριστώ. Η Σοφή Ιντεβέλντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη. Δεν ε, με καθησυχάσατε, ούτε κι εσείς. Είναι περίπλοκο το ζήτημα ε, για την εποπτεία μπορεί να έχουμε σωστούς κανόνες, καλούς κανόνες, ενισχύει, όμως το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων διαφεύγουν του ελέγχου για διάφορους λόγους. Έναν τον αναφέραμε, διότι υπάρχει διασυνοριακή διάσταση, Φερρυπίν. Επίσης, ε, αυτό που κάνουν θεωρείται τουλάχιστον από τις ίδιες υπηρεσίες πληροφοριών, ε, ως επιτοπλίστων σύνομο. Ακόμη και το πρόγραμμα βασανιστήριων της CIA ε, τρόπον την είχε λάβει έγκριση. Υπήρχαν ε, ε, νομικού περιεχομένου διαταγές που νομιμοποιούσαν τη δράση τους. Μπορεί τότε να λέγαμε ότι είναι ανήθικο και απάνθρωπο, αλλά αυτό γινόταν. Ε, στην η ιστορία της DCHQ ε, σε Ολλανδική, στην Ολλανδική επικράτεια ε, ε, καταλαβαίνετε ότι πάλι θεωρήθηκε ότι κινούνταν μέσα στα περιφέρεια του νόμου υπηρεσίας πληροφοριών. Και από διαβάζουμε στις εφημερίδες, ένας Αυστριακός βουλευτής είπε ότι η BND κατόπιν αιτήματος του, της NSA ε, κατασκόπευε Ολλανδικές υπηρεσίες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πώς είναι δυνατόν να υπάρξει έλεγχος σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Και ε, νομίζω ότι οι προηγούμενοι ομιλητές, οι ομιλητές του προηγούμενου πάνελ θα συμφωνήσουν με τις ανησυχίες μου από τη διαστολή με αυτά που μας είπατε εσείς. Και λέτε να πάνε στα δικαστήρια, μα τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν ότι παρακολουθούνται στα πλαίσια μιας τέτοιας μαζικής ε, παρακολούθησης. Ή τι, ε, να πάει το δικαστήριο και να τους πει ή οποιοδήποτε θεσμός να, να τους πει λοιπόν δεν μας αρέσει που μας κατασκοπεύετε. Δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει, χρειάζεται ένα κρατεότερο σύστημα ελέγχου Ξέρουμε ότι τα εφιστάμινα συστήματα έχουν αποτύχει. Δείτε τι έγινε με τα προγράμματα της CIA, με την κατασκοπία από πλευράς ε, ε τη CIA, το, την TCHQ, ε, την ε, η κυβερνητική υπηρεσία, το αρχηγείο δηλαδή της κυβερνητικής υπηρεσίας ε, πληροφορία. Βλέπουμε ότι κάποιε επιχειρήσει ε, πραγματικά διαφεύγουν οποιοδήποτε ελέγχου. Σα ευχαριστούμε, λέει ο κύριο Μωρέ, ο κύριο Στρέμπελε από πλευρά του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Yeah. <clears throat> Ich Να επισημάνω ότι εμεί οι βουλευτές μπορούμε να ελέγχουμε μόνο αυτά που μαθαίνουμε, αυτά που μα γνωστοποιούνται και βεβαίως αυτά που κατανοούμε. Φυσικά δεν είμαστε κανείς μας ε, εμπειρογνώμονες όσον αφορά τις ε, μυστικές ε, υπηρεσίες. Και αυτό το λόγο χρειαζόμαστε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη Γερμανία υποστήριξη από εμπειρογνώμονες, από ειδικού. Υπάρχει η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από εννέα βουλευτές αλλά η Επιτροπή αυτή προσπαθεί να βρει συνεργάτες από διάφορους τομείς πρόκειται δηλαδή για ένα μείγμα μεταξύ εμπειρογνωμοσύνης την οποία αποκτούμε μέσω της συνεργασίας μας με ε, εξωτερικούς συνεργάτες και ε, αφετέρου κοινοβουλευτικού ελέγχου και γι' αυτό το πρότυπό μας είναι το Κογκρέσο των ΗΠΑ, όπου οι βουλευτές, 60 τον αριθμό, έχουν το δικαίωμα προσβά... πρόσβασης στις μυστικές υπηρεσίες για να μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα ελέγχου τους. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω και το ανέφερε και η Ολλανδή συνάδελφος αλλά και ο Αυστριακός συνάδελφος και είναι το εξής. Επιτρέπεται παράνομα μυστικά να παραμένουν μυστικά. Επιτρέπεται οι κυβερνήσεις που έχουν ε, λάβει με παράνομο τρόπο πληροφορίες να τις διατηρούν μυστικές. Είναι, επιτρέπεται να παρακολουθούνται ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιτρέπεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας να αποκρύπτει τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες και η απάντηση είναι σαφής. Παράνομα αποκτηθήσεις πληροφορίες δεν επιτρέπεται να παραμένουν μυστικές αλλά θα πρέπει να διατίθενται στην ε, διάθεση, να τίθενται στη διάθεση ε, των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Και κάτι ακόμη. Ε, οι αποκαλύψεις Snowden αποτέλεσαν μια τομή, διότι έκτοτε γνωρίζουμε πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε στο παρελθόν. Δεν θα πρέπει λοιπόν να βγάλουμε το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία ότι χρειαζόμαστε μια ε, ευρωπαϊκή ρύθμιση για τους πληροφοριοδότες. Για πληροφοριοδότες δηλαδή που αποκαλύπτουν υποθέσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι μόνο στη ΣΥΠΑ, ώστε αυτοί οι πληροφοριοδότες, άνθρωποι δηλαδή μέσα από τις μυστικές υπηρεσίες, να μπορούν να ενημερώνουν και το κοινό και την κοινή γνώμη δηλαδή και, τους και, τα κοινοβούλια και τους βουλευτές είτε πρόκειται για επιχειρηματικά μυστικά ε, ε, όπου ενδεχομένως έχουν υπάρξει σκάνδαλα. Αλλά χρειαζόμαστε αντίστοιχες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα εκείνων των ανθρώπων που αποκαλύπτουν τέτοιου είδους πληροφορίες όπως έκανε ο Έντουαρτ Σνόντεν. Δηλαδή να διασφαλίζουμε και να εξασφαλίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα φυλακιστούν, δεν θα καταλήξουν στη φυλακή. Τέτοιου είδους κανόνες, τέτοιου είδους νομικές διατάξεις χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Λοιπόν, έχουμε ε, στενά περιθώρια χρονικά σε μισή ώρα θα πάμε για μεσημεριανό. Θέλω να θα δώσω την ε, δυνατότητα και στους ομιλητές να απαντήσουν. Έχουμε λοιπόν ε, ξαφνικά ε, πάρα πολλούς ομιλητές, πάρα πολλές ερωτήσεις και θα ήθελα να περιορίσουμε ο καθένας μας τις παρεσβάσεις του στο, σε ένα-δύο λεπτά αν γίνεται. Ξέρω ε, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για τις τοποθετήσεις των βουλευτών, αλλά ε, δεν ξέρω τι γίνεται και σε άλλες χώρες. Αν το, κάνει αυτός, αν το κάνουμε αυτό εδώ δεν πρόκειται να ακούσουμε καμία ε, ερώτηση. Ε, ίσως θα μπορούσαμε δηλαδή σε μια τέτοια περίπτωση να φτάσουμε μέχρι αύριο το πρωί. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Γερμανία, αν υπάρχει εκεί χρόνος όμως. Εσείς είστε Σκοτσέζος, δεν ξέρω αν εκεί έχετε όρια για το χρόνο ομιλίας. Τέλος πάντων, ας πούμε τώρα δύο λεπτά και ας δούμε πώς θα πάει. Ξεκινούμε με τον συντονιστή του ΕΛΚ από τη Γερμανία. Βλέπω εδώ την ε, Μόνικα, την κυρία Γολμάιερ. Η Μόνικα Ολμαϊρ έχει το λόγο. Συντονιστής για το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Θα τα καταφέρω σε δύο λεπτά. Ούκεν το πόλο το F. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ε, σωστό ε, οι βουλευτές να λαμβάνουν εμπειρογνωμοσύνη μέσα της συνεργασίας τους με εξωτερικούς συνεργάτες. Και είναι σαφές αυτό και είναι και γνωστό. Δεν μπορεί κάθε βουλευτής θα ήταν μια υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του ε, να θεωρήσουμε ότι κάθε βουλευτής ε, γνωρίζει σε βάθος ε, τα ζητήματα που σχετίζονται με τις μυστικές υπηρεσίες. Υπάρχουν εμπειρογνώμονες, υπάρχουν ειδικοί και βεβαίως μπορούμε να έχουμε την, απότηση, την απέτηση να ε, μας ενημερώνουν εκείνοι. Κύριε Στρόμπελε, μιλήσατε για, τα, για, τις, μυστικές, για τις παράνομες πληροφορίες. Εγώ θα έθετα το ερώτημα πώς ακριβώς θα αξιολογηθεί αυτός ο παράνομος χαρακτήρας και ταυτόχρονα θα, μπορούσα, θα, έπρεπε, θα ήθελα και να επισημάνω ότι για παράδειγμα στα ζητήματα της βίας ή των βασανιστήριων νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα ε, υποστήριζε αυτού του είδους τις μεθόδους αλλά υπάρχει μια ομόφωνη, ε, μια ε, κοινή στάση ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι, μέθοδο, αυτές οι μέθοδοι. Επίσης, χρειαζόμαστε διαφάνεια. Και για να διασφαλιστεί διαφάνεια θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που μας διαβιβάζονται δεν θα καταλήξουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να δημιουργηθούν κίνδυνοι και για τη ζωή ανθρώπων. Άρα θα πρέπει να ε, ορίσουμε και ποιες θα είναι οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε βουλευτές που δεν θα τηρούν τους κανόνες. Όσον αφορά τους πληροφοριοδότες, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιους πληροφοριοδότες, αλλά δεν είναι και σωστό να τους εκθιάζουμε. Ε, θα πρέπει βεβαίως να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που θα προστατεύει τους ανθρώπους που δίνουν πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και να είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να διαρρέουν πληροφορίες ε, προς τα έξω να μην δημοσιοποιούνται πληροφορίες οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για ανθρώπους και νομίζω ότι ε, οι πληροφορίες που λάβαμε για το ε, NSA ε, πράγματι αποδείχθηκε ότι πολλές από αυτές τις αποκαλύψεις ε, μας ε, χρησιμεύσαν και στη διαλεύκανση ε, υποθέσεων και στην αποτροπή επιθέσεων. Πάντως σε κάθε περίπτωση η προσέγγιση που θα πρέπει να υιοθετήσουμε θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένη κατά περίπτωση δηλαδή. Ευχαριστώ Μόνικα. Από την ε, Αυστριακή Βουλή ο κύριος Πέτερ Μπίλς. Okay. Ich lerne gerade Knöpfe zu Αχ, μόλις τώρα μαθαίνω να ε, λειτουργώ αυτά τα κουμπιά. Η συνάδελφος από τις κάτω χώρες ε, ε, με ανέφερε πριν. Είμαι ο βουλευτής που δημοσιεύει συστηματικά έγγραφα της NSA και του BND της Γερμανίας. Ο κύριο Στρόμπελ ανέφερε ήδη το πρόβλημα στο οποίο θέλω να αναφερθώ και εγώ. Μέρος των μυστικών υπηρεσιών του έργου τους είναι ε, ε, παράνομο με βάση την νομοθεσία. Το ότι εγώ ως βουλευτής πρέπει να λάβω τέτοιου είδους έγγραφα που διέρευσαν από την NSA το βρίσκω απαράδεκτο. Θα πρέπει δηλαδή να διακρίνουμε μεταξύ εγκληματικών ενεργειών της NSA και του BND μέσω μιας συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που προφανώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Να αφήσω στην άκρη προς το παρόν την υπόθεση NSA και να σας επισημάνω ε, ένα άλλο πρόβλημα. Διαπιστώσαμε στην Αυστρία ότι η αντιτρομοκρατία, η ε, αντικατασκοπία δεν ε, λειτουργεί σωστά. Και μάλιστα συνεργάζεται στενά με τις μυστικές υπηρεσίες. Ελέγχω εδώ και 30 χρόνια αυτού του είδους της δραστηριότητας και βλέπω ότι σε διεθνώς ε, επίπεδο έχει δημιουργηθεί κάτι σαν μια οικογένεια. και υπάρχει ένας μεγάλος αδερφός στην Ουάσιγκτον, ένας μεσαίος αδερφός στο Βερολίνο και ένας μικρός αδερφός στη Βιέννη. Και σε πολλές περιπτώσεις ε, ε, αποδεικνύεται ότι ο μικρός αδερφός δεν πρόκειται να ελέγξει παράνομες δραστηριότητες των, του, του μεγάλου ή του μεσαίου ε, αδερφού. Αυτή ακριβώς είναι η του μεσαιου αδερφου αυτη ακριβως ειναι η κατασταση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Αυστρία. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε όχι μόνο τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την συνεργασία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά μήπως θα έπρεπε σε κάθε χώρα να διαχωρίσουμε τις υπηρεσίες αντικατασκοπίας από τις μυστικές υπηρεσίες μας σε κάθε χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ιταλία, η κυρία Κατρίνα Τσινίτσι, Ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συζητητές που συμμετέσχουν και του πρώτου πάνελ που ήρθαν στην ε, συνάντησή μας και μας είπαν πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, όλες τις χώρες. Όταν μιλούμε για υπηρεσία πληροφοριών, μιλούμε για ασφάλεια στις χώρες μας. Η ασφάλεια απαιτεί κάποιες παρεμβάσεις. Βεβαίω όμως το θέμα άπτεται των ατομικών δικαιωμάτων και του ιδιωτικού βίου. Άρα αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει για αυτή τη σημαντική δραστηριότητα είναι να υπάρξει μια δραστηριότητα δημοκρατικού ελέγχου. Που τέτοιο θα πρέπει να συγκροτηθεί. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε ο καθηγητή Κάμερον για το Κοινοβουλίο. Επίση χρειάζεται και έλεγχο από κάποιε ειδικέ επιτροπέ, ειδικού φορεί. Πρέπει φυσικά να συμμετέχει και κάποιο ε, δικαστή που να έχει κατάρτιση ανάλογη και θα συμβαίνει πάρα πολύ στην ε, προστασία των δικαιωμάτων. Πάντως, συνήθως οι υπηρεσίες πληροφοριών ασχολούνται με πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Πολλές φορές πρόκειται για εγκληματική δραστηριότητα. Πολλές φορές είναι το θέμα διασυνοριακό. Οπότε και οι συνέπειες αφορούν περισσότερες χώρες. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι συντονισμός και όχι μόνο για τις υπηρεσίες πληροφοριών συντονισμός και για τους εποπτικούς φορείς. Άρα τι να κάνουμε, τι πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ πέστε μου, θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό να γίνει επί τη βάση της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. αυτά τα οποία προβλέπει η Σύμβαση των Δικαιωμάτων θα μπορούσαν να είναι βάση για να προκύψει κάτι το οποίο να είναι αφετηρία, πρόβλεψη αυτού του δημοκρατικού ελέγχου που να είναι και νομικά κατοχυρωμένος και αποτελεσματικός. Γιατί όπως λέγαμε μιλούμε για κάποια εγκλήματα τα οποία απασχολούν τις υπηρεσίες πληροφοριών. Και πολλές φορές η δραστηριότητα αυτή των υπηρεσιών εμπλέκει περισσότερες χώρες. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Κατερίνα. Και όπως πρέπει, να να συνάδελφος από τα Αθηνικά Κοινοβούλια. Πρόκειται από την Πορτογαλία. Είναι ο Πρόεδρος του Εποπτικού Φορέα, Φερνάντο Νεκρά. Φερνάντο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο ε, για να συμφωνήσω και με τον κύριο Σάντες από την Ισπανική Βουλή. Θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικός είναι ο κοινοβουλευτικό έλεγχο ε, και ο πολιτικό έλεγχο. Ε, ξέρετε, στα κοινοβούλια εκπροσωπούνται τα διαφορετικά οράματα των πολιτών, οι διαφορετικές θεωρήσεις ως προς την ασφάλεια και ως προς την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ε, οπότε δεν μπορεί παρά να ασχοληθούμε και με το τεχνικό κομμάτι και μπορούμε να λειτουργήσουμε με ε, ελεγκτικές επιτροπές όπου συμμετέχουν και δικαστές και βουλευτές αλλά και τεχνικοί που θα λογοδοτούν όμως ε, στη Βουλή και ένα, μια τέτοια μεικτή επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα και από τεχνικής και από πολιτικής πλευράς να δώσει την προσφορότερη απάντηση στα προβλήματα που ε, δημιουργούνται ε, σε σχέση με την ασφάλεια κατά τη λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν τόσο σύντομος. Ο κύριος Στούτσε ε, το είπατε τελευταία στιγμή, μπορείτε να είστε σύντομο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο κύριο Στούκη. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θα ήθελα τη γνώμη σα για μια δραστηριότητα αφεντικού έλεγχου από πλευρά τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Πώ να τον έχουμε συγκεκριμένε πληροφορίε για κάποια συγκεκριμένα προβλήματα ή πληροφορίε δημιουργούνται κατά τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις προέρχονται από υπηρεσίες. Υπηρεσίες πολλές φορές άλλων χωρών. Ποια είναι η πηγή τέτοιων πληροφοριών, ποιος βρίσκεται πίσω από την παροχή αυτών των πληροφοριών, γιατί εδώ έχουμε δραστηριότητε που θα πρέπει να επιδέχονται και να υπόκεινται σε έλεγχο και να αποφύγουμε παραβάσεις του δικαίου. Για πέστε μου πάνω σε αυτή τη γνώμη σας. Thank Ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστώ που ήσασταν τόσο επιθαρχημένοι και δεν υπερβήκατε το χρόνο που σας αναλογούσε. Θέλω να ε, σας καλέσω να δείτε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Η κυρία Χολμάγερ μας μίλησε για αυτό το σημαντικότατο και δύσκολο πρόβλημα. Θυμηθείτε ότι ε, ήταν πολύ ευαίσθητα τα ζητήματα και καταφέραμε μετά από συνεργασία των πολιτικών ομάδων σε κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Παρακαλώ, σας παραπέμπω ε, να διαβάσετε το ψήφισμα αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Δίνω το λόγο αμέσως στον καθηγητή Κάμερον για να απαντήσει σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις. Ε, και μου αρέσει γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν, υπηρεσίες πληροφοριών, αστυνομία, για όλα αυτά τα σχετικά ερωτήματα, όσοι ενδιαφέρονται να διαβάσουν παρακαλώ την έκθεση 2007 για την Επιτροπή, ε, της Επιτροπής Βενετίας, ε, γιατί εκεί μιλάμε για τις εσωτερικές ε, ε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και Έχουμε κάνει υπό μακροσκελέστατες και ε, βαρετές συζητήσεις γι' αυτό, αλλά δεν σας ε, λέω να παρακολουθείτε αυτές. Σας παραπέμπω στην έκθεση του 2007, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και έχει πολύ σημαντικά στοιχεία. Όπως ε, λένε οι Αμερικανοί, κάντε τους υπολογισμούς για να βρείτε την απάντηση. Do the math. Αν έχετε μια μεγάλη υπηρεσία πληροφοριών, ε, δεν μπορείτε να έχετε μια μικροσκοπική ελεγκτική ομάδα για μια πελώρια τεράστια ε, ε, ε υπηρεσία πληροφοριών. Είναι απλά τα πράγματα. Ε, υπάρχει μια μόνιμη ομάδα που παρακολουθεί την ε, Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών παραδείγματο χάρη, την παρακολουθεί όλη την ημέρα, κάθε μέρα ε, και δεν χρειάζεται να είναι στο ίδιο κτίριο, αλλά μπας και την παρακολουθεί διαρκώς. Υπάρχει και ένα επίπεδο παρανόηση σε σχέση με αυτό που προσπαθώ να πω εδώ για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μπορώ να σας πω ότι Καταλαβαίνω την ευαισθησία που έχουν οι συνάδελφοι από την Ισπανική και την Πορτογαλική Βουλή για αυτό το ζήτημα, διότι αγωνίστηκαν ε, για την, το δημοκρατικό έλεγχο και για τον έλεγχο ολόκληρη τη διοίκηση ε, και του κυβερνητικού μηχανισμού και έρχεται κάποιο και του λέει τώρα δεν μπορείτε. Όχι, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ λεπτό αυτό το ζήτημα και δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο. Απλώ έλεγα πω υπάρχουν ε, διαφορετικά μοντέλα και ταιριάζουν σε κάποια κράτη-μέλη. Απλώς σας είπα ότι για την στρατηγική συλλογή πληροφοριών, δηλαδή την, ε, τις πληροφορίες σημάτων, ε, δεν είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος αυτός. Υπάρχουν όμως εναλλακτικέ λύσεις. Ποιες είναι αυτές. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται ένα υβριδικό σώμα, ένα υβριδικό φορέα όπως συμμετέχουν και οι δικαστέ. Πρώην βουλευτέ μπορεί να μετάσχουν ή και ενεργοί, αλλά αυτό είναι λίγο πιο προβληματικό και αυτοί οι βουλευτέ μπορούν να ε, διοριστούν από το κοινοβούλιο, να υπάρχει λογοδοσία παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν τρόποι δηλαδή να συνδεθεί ε, το κοινοβούλιο με αυτό το ελεγκτικό σώμα και μπορεί να μου αντιτάξετε α, ε, εντάξει τι νομοθετούμε για τους πυρηνικούς αντιδραστήρες αυτό το κατέχουμε το ζήτημα βεβαίως αυτός είναι ο ρόλος του κοινοβουλίου ε, προσφεύγει σε εξωτερική πραγματογνωμοσύνη το συζητεί και νομοθετεί αυτή είναι η δουλειά των ε, ε, κοινοβουλίων γιατί μόνο εκείνα νομιμοποιούνται. Δεν πάτε όμως να ελέγξετε και τον πυρηνικό αντιδραστήριο να δείτε αν έχει... Ε, ε, υπάρχουν ε, ναι. που θέτουν εν κινδύνο την ασφαλή λειτουργία του, του συστήματος. Ε, αυτό ε, σας είπα. Υπάρχουν τρόποι να συνδεθεί η νομιμοποίηση του Κοινοβουλίου, η αποκλειστική νομιμοποίηση του Κοινοβουλίου με αυτόν τον ελεγκτικό σώμα, γιατί σας λέω ότι δεν υπάρχει τεχνική πραγματογνωμοσύνη, τόσο ώστε σε κάθε λεπτομέρεια και με πάγιο τρόπο να ελέγχει το Κοινοβούλιο. Αυτό είπα μόνο για να μην υπάρξει παρανόηση. Κοιτάξτε, ε, ας περάσω στο επόμενο ερώτημα. Και οι ίδιοι οι πολίτες μας μπορεί να θυμιστούν απειλή, ε, ε, οπότε, ξέρετε, έχει γίνει όλη τη συζήτηση για τους foreign fighters, τους ξένους μαχητές, και ένα πράγμα που κάνουμε είναι για να απομακρύνετε τα στοιχεία για τους υπηκόου υπηκόους από τα δεδομένα που μεταβιβάζετε σε τρίτες χώρες. Ναι, όμως θα μεταφέρεται δεδομένα άλλων υπηκών, άλλων κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Σουηδία που έπαιρνε τα στοιχεία κάποιων και τα έστελνε στη ΣΥΠΑ, γιατί ήταν για Φινλανδούς ή για Αυστριακούς, ας πούμε. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι το βασικό μέλημα είναι να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των υπηκών όλων των κρατών μέλων. Αυτό πρέπει νομοθετικά να κατοχυρωθεί. Όχι να απαγορευτεί, να πούμε, ε, σκεφτείτε το σοβαρά πρωτού ε, μεταβιβάσετε στοιχεία που αφορούν υπηκός άλλων χωρών. Τώρα για την υποδοχή, την πρόσληψη στοιχείων από άλλους μπορεί να γίνει ανάλυση μόνο αν πληρούνται τα κριτήρια που ούτως ή άλλως ε, προβλέπονται ε, στο κανονισμό σας, δηλαδή αν ήταν να τα συλλέξετε εσείς οι ίδιοι. Αλλά μην ξεχνούμε ότι ε, δικαιώματα για την ιδιωτική ζωή έχουν και οι αλλοδαποί και οι μη μόνιμα διαμένοντες. Ε, σας, σας παραπέμπω και πάλι στην έκθεση του 2015. Είναι, ε, ε, ε, ε συμπεριλαμβάνει περιστατωμένα στοιχεία για τις πληροφορίες σημάτων Και εκεί βλέπουμε ότι για το πρόγραμμα της CIA e, που είναι ντροπή και όνειδος για κάθε δημοκρατική κοινωνία συνδέεται με το ζήτημα της εποπτείας από ποια πλευρά ότι παρακάμφθηκε ο έλεγχος. Δείτε από πλευράς ε, της γερουσίας ε, ε, τον ήπα. υπήρχε ένα σύστημα, αναφέρεται μέσα στην έκθεση, αλλά η θελημένα παρακάμφθηκε μετά από πολιτική πίεση. Αυτό ήταν το πρόβλημα με τις διαρροές που προ... έγιναν στον τύπο από τους αξιωματούχους ε, της CIA. Δεν το δικαιολογώ, δεν το δικαιολογώ καθόλου σε καμία περίπτωση. Απλώς σας είπα για πώς ξέσπασε το σκάνδαλο. Για την NSA τι έγινε. Οι πληροφορίε σημάτων δεν θεωρήθηκε ότι επηρεάζουν κατά τον ίδιο τρόπο την ιδιωτικότητα Υπάρχει μία μεγαλύτερη αποδοχή. Δηλαδή λένε άμα εμείς δεν ε, παραβιάζουμε την ιδιωτική σας ζωή, βλέπουμε αν ε, ε, έχετε εσείς σχέση με όπλα μαζικής καταστροφής, χημικά όπλα, βιολογικά όπλα κτλ. Όμως υπάρχει μία επίγνωση ότι ε, αυτό δεν ισχύει ε, και γι' αυτό ε, πέρασε η νομοθεσία στη ΣΥΠΑ, διότι τα περί εποπτείας δεν έφταναν. Το, το διαπίστωσε αυτό η γερουσία των ΗΠΑ και αν δείτε τι συμβαίνει στη ΣΥΠΑ είναι κατακαιρματισμένη και αναποτελεσματική υπηρεσία. Υπάρχουν κάποιοι πολύ καλοί στο προσωπικό, όμως δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο θα ελπίζαμε και υπάρχουν πολύ και διαφορετικοί λόγοι ε, για αυτό και αναφέρονται επακριβέστατα μέσα στην έκθεση Επιτροπής Βενετίας. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο να λογοδοτούν και οι υπουργοί. Οι υπουργοί όμως πάντοτε έχουν τη δυνατότητα να κρύβονται πίσω από το απόρριτο. Και σε αυτό εγγύεται και μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η NSA. Dr. please go ahead. Thank you, Chair. Uh, Ευχαριστώ. Uh, uh, ο κύριος Ετχάιμερ, σας ευχαριστώ ε, για τις ε, ερωτήσεις σας. Τρία να σας αναφέρω. Και συγγνώμη δεν καλύψω όλες τις ερωτήσεις, αλλά νομίζω ότι ο καθηγητής Κάμερον ήδη κάποιες τις κάλυψε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για την σχέση μεταξύ των διοικητικών αρχών και των υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτό δεν θα το δείξει η έκθεση της κοινωνικής υπηρεσίας ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και ο λόγος είναι ότι η σχέση μεταξύ αυτών των φορέων δεν προβλέπεται κατά κάποιο τρόπο από το δίκαιο. Οι σχέσεις αλλά και οι συναλλαγές του στο ΣΥΠΗΝ δεν είναι κάτι που διέπεται ή ρυθμίζεται από τον νόμο. Αυτό είναι το θέμα και ακριβώς αυτό είναι το συμπέρασμα το οποίο θα μπορούσαμε να εξαγάγουμε από τη σχέση μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών πληροφοριών. Ούτε αυτό ρυθμίζεται από το δίκαιο. Σε κάποια κρατημέλη ορίζεται σαφώς ότι όλα αυτά είναι άκρος απόρριτα και δεν θα πρέπει να διέπονται από νομική ρύθμιση. Οπότε Οπότε επομένω και η Εθνική Υποτική Αρχή θα έπρεπε να είναι εις θέση να εξετάσει τουλάχιστον την κατάληξη της διαδρομής των πληροφοριών τόσο ώστε να μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι ούτω ώστε να προστατευτούν τα ατομικά δικαιώματα. Πριν αξιοποιηθεί η πληροφορία. Τώρα κάποια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση είχαμε. Αφορούσε το αυτό το οποίο έγινε, το οποίο κάνουμε, ή να επιτρέπεται από το νόμο και ποιες είναι οι δυναμίες του συστήματος σε αυτή τη φάση δεν θα έδινα σημασία σε αυτό, στα, στα τροτά της εποπτείας. Να μια ματιά στα εθνικά δίκαια. Αυτό που θα έκανα θα ήταν να δω τι προβλέπει ο νόμος. Συμφωνώ μαζί σας ότι χρειάζεται να υπάρχει ευελιξία και έτσι οι υπηρεσίες να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Όμως, προσπάθησα να σας πω και στην εισήγησή μου ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ορισμός, κάποια περιχαράκωση για να καταλάβουμε ποια είναι η εντολή της υπηρεσίας και μέχρι που μπορεί να φτάσει. Άρα, θα πρέπει ξανά να δούμε τι προβλέπει το δίκαιο. Και κάποιες ε, χώρες κάνουν μεταρρυθμίσεις του σχετικούς νόμους να προσπαθήσουν να δουν πώς θα υπάρχει ταυτόχρονα και διαφάνεια και ευελιξία. Ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον το συμπέρασμα του κ. Μπίκφορντ προηγουμένω που έλεγε ότι κάποια κράτη μελέφθασαν στο επίπεδο τη απόφαση Λεάνδρου και όχι τη απόφαση Κλάς. Εγώ δεν είμαι πεπισμένο ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και βέβαια μιλάω για τι πρώιμε φάσει τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, αλλά λέω τώρα για το κατά πόσο πρέπει να υπάρχει κάποια διαφάνεια ε, από πλευρά νομική και κατά πόσο υπάρχει αυτή η διαφάνεια λοιπόν σε κάποια κράτη μέλη. Ο Πρόεδρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάρα πολύ που μα ενημερώσατε, συναδελφοί. Ευχαριστώ που ήρθατε. Και ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην συνάντηση. Τώρα έχουμε κάποιες ε, ανακοινώσεις από πλευρά μου δυόμιση θα ξαναρχίσουμε για να εμβαθύνουμε περαιτέρω σε αυτά τα θέματα και σας υπενθυμίσω σε όλους ότι τα εργαστήρια θα γίνουν με τέτοιο τρόπο που θα μπορέσετε να τοποθετηθείτε, να πείτε την ελεύθερη άποψή σα, να μας πείτε τις εμπειρίες του καθημερινού κοινοβουλευτικού βίου που περνάτε. Επίσης έχουμε τους συνοδούς των αντιπροσωπιών και έχουμε συνάντηση αυτού του προσωπικού μεταξύ 2 και 2,5 στο 4Q1 αυτού του κτηρίου. Πρόκειται για το προσωπικό που συνοδεύει τους ε, εθνικούς βουλευτές. Είναι μια συνάντηση που προβλέπεται για σας. Μεταξύ 2 και 2,5 όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες ας ρωτήσει το τη γραμματεία μας. Άρα, όλα αυτά αφορούν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των, ε, των προσπαθειών μεταρρύθμισης των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών. Οπότε παρακαλώ να συναντηθείτε όλοι εδώ στις 2.30 ακριβώς για να συνεχίσουμε. A good break until then, but please don't... Καλή όρεξη και μην αργήσετε. 2.30, 2.30 ξαναλέω ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ για τόσο ενδιαφέροντα συνεδρία. 2.30.